Καλημέρα σας, λέει ο πρόεδρος. Είστε έτοιμοι? Αρχίζουμε την συνεδρίασή μας. Και πριν... To read um, out uh, a letter I got from the interpreters. Um, so I'll do that on their behalf. Uh, Έχουμε κάτι από τους διερμηνείς. Να σας το πω εκ μέρους τους. Οι διερμηνείς ε, δυστυχώς πρέπει να σας ενημερώσουν ότι υπάρχει μια εργασιακή διαφορά ε, και η οποία συνεχίζεται ως προς τη διοίκηση του Κοινοβουλίου για νέες συνδίκες εργασίας τους και επομένως η ποιότητα της δερμηνίας ε, κινδυνεύει και γι' αυτό λυπούνται αλλά πρέπει να σας ενημερώσουν ότι θα σταματήσουν να εργάζονται ακριβώς στις 6 ώρα την ώρα που προβλέπεται η λήξη της συνεδρίας. Αυτά από πλευρά των Δερμήνιων Και τώρα πάμε στην ε, ημερησία διάταξη της συνεδρίασης. Έχουμε κάποιες ε, μελέτες πολύ ενδιαφέροντος που έχουμε στα χέρια μας εδώ στην, στο πλαίσιο της Επιτροπής μας, τάξ 3. Και σήμερα έχουμε ένα εργαστήριο που αφορά την ε, φορολογία και καταπολέμηση νομίζεις εσόδων με τα κρυπτονομίσματα ψηφιοποίηση και ευρωπαϊκό εξάμεινο και έχουμε δύο μελέτες προς ε, παρουσίαση. Ε, αυτοί που συνέταξαν τις μελέτες. Πρώτα-πρώτα έχουμε τον καθηγητή Χούμπεν από το Πανεπιστήμιο της ε, Αμβέρσας και θα μας πει τα του νομικού πλαισίου για τα κρυπτονομίσματα, για το ξύλιμα νομίσματος σε σχέση με το κοινοτικό δίκαιο και εδώ θα τονιστούν ε, οι βασικοί στόχοι των αρχών δηλαδή να υπάρχει κάποιο είδου κοινή πολιτική, κοινέ πολιτικές ούτως ώστε να καταπολεμηθούν οι παράνομες δραστηριότητες και πρακτικές όσον αφορά το οικονομικό έγκλημα, το ξέπλυμα χρήματος και την φοροδιαφυγή. Βέβαια, η, φο... η επιβολή φορολογίας στην ψηφιακή οικονομία είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πολιτικά και οικονομικά. Θα πρέπει επίσης το πλαίσιο της φορολογικής πολιτικής να το προσαρμόσουμε στην σημερινή πραγματικότητα. Η κυρία Χατζίεβα, ε, αν λέω καλά το όνομά της, είναι η ιδρύτρια και διευθύντρια του φορέα Διάλογος για την Ευρώπη. Θα μας πει δύο λόγια για κάποια μελέτη που έχει ετοιμάσει για την Επιτροπή Τάξη 2. Επίσης έχουμε τον καθηγητή Βέλα εδώ από την ε, Οξφόρδη, από το Πανεπιστήμιο. Ε, ασχολείται με το κέντρο ε, φορολόγησης των επιχειρήσεων και θα μας πει τι διεθνείς εξελίξεις έχουμε, τι μέσα, ε, πάντων τι μέτρα μάλλον έχουν θεσπιστεί για αυτό το μέτωπο. Ε, επίσης θα ολοκληρώσουμε όσον αφορά την ε, φορολογία, πώς θα αντιμετωπιστεί κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Κύριο Βαλέρ Μουταρλίε είναι διευθυντή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρότεινε να μα πει για το τι γίνεται όσον αφορά ε, αυτές τις ε, φορολογικές τακτικές ε, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και για το τι γίνεται με τις πολυεθνικές που ακριβώς ακολουθούν τέτοιες τακτικές προκειμένου να γλιτώσουν φόρους. Κύριε Χούμπεν, καθηγητά στο Πανεπιστήμιο της ε, Αμβέρσας, παρακαλώ μπορείτε να αρχίσετε να μας κάνετε την παρουσίασή σας για 15 λεπτά κατόπιν θα έχουμε ερωταπαντήσεις με τα μέλη της ε, Διερευνητικής Επιτροπής. Χούμπεν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε για την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σε σχέση με τη μελέτη μας όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα και το blockchain. Καθώς ε, και το σχετικό νομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά το οικονομικό έγκλημα και την ε, το ξέπλυμα οικονομικού χρήματο. Όλο ε, και περισσότεροι νομοθέτε ανησυχούν σχετικά με του αγκληματίε οι οποίοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερα τα κρυπτονομίσματα για παράνομε δραστηριότητε όπω το ξέπλυμα βρωμικού χρήματο, η χρηματοδότηση τη τρομοκρατία και η φοροδιαφυγή. Και το πρόβλημα είναι σημαντικό. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ακριβώ το μέγεθό του, αλλά υπάρχουν εκθέσει που εκτιμούν ε, πω ανέρχεται σε 7 δισεκατομμύρια ευρώ ανά τον κόσμο. Ε, και η μελέτη μας εξετάζει αυτό το φαινόμενο από, νομική, από τη νομική πτυχή, δηλαδή τη χρήση ε, των κρυπτονομισμάτων για αυτούς τους σκοπούς, το ξέπλυμα χρήματος, ε, την τρομοκρατία και άλλα ζητήματα. Ο συνάδελφος θα κάνει μια παρουσίαση ως προς τα κύρια ζητήματα και στη συνέχεια θα σας αναφέρω τα πορίσματα της μελέτης μας. Αυτό που κάναμε είναι το να εξετάσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά ε, αυτής της αγοράς και να δούμε πώς ακριβώς διαμορφώνεται αυτή η αγορά, ποιοι είναι οι βασικοί παίκτες σε αυτά τα συστήματα κρυπτονομισμάτων και τι ακριβώς συμβαίνει με το ε, bitcoin και τα bitcoin σε εκείνα, ε, τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στην αγορά. Και από εκεί και μετά έχω, εξετάζουμε το πώς ακριβώς ε, σχετίζονται με την, ε, και με την τέταρτη οδηγία για την καταπολέμηση του ξυλίματος του βρώμικου, ε, βρώμικου χρήματος αλλά και τα ζητήματα της φοροδιαφυγής και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Και σε συνέχεια της εξέταση που κάναμε τη αγορά των κρυπτονομισμάτων, εξετάσαμε την αποτελεσματικότητα του νομοθετικού πλαισίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση των κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιούνται για αυτού του παράνομου σκοπού. Και το κάναμε, κάναμε την αξιολόγηση με βάση μία σειρά από ερωτήματα. Καταρχήν, είδαμε το κατά πόσο ο ορισμός ε, αυτών των κονικών νομισματών όπως λέγονται ε, είναι επαρκής όπως αυτός περιλαμβάνεται στην οδηγία. Και από εκεί και μετά εξετάζουμε ε, το κατά πόσο εκείνοι οι οποίοι εκδίδουν τα κρυπτονομίσματα περιλαμβάνονται στην ειδική κατηγορία των ενεχόμενων οντοτήτων. Και από εκεί και μετά θέσαμε το ερώτημα το κατά πόσο ε, πράγματι τίθεται υπό την επαρκή εξέταση χρήστες των κρυπτονομισμάτων. Ε, και εδώ βασιζόμαστε στην οδηγία σε ό,τι αφορά το cash control και την οδηγία για τον έλεγχο των μεταφορών, έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο καλύπτονται και μεταφορές κρυπτονομισμάτων. Επίση, είδαμε κατά πόσο υπάρχει ανάγκη για να υπάρξει ε, μια πιο περιεκτική προσέγγιση, μια πιο ευρεία προσέγγιση που θα ε, προποθέτει άδειε για τα κρυπτονομίσματα. Ε, και για παράδειγμα θέσαμε το ερώτημα του κατά πόσο θα έπρεπε να θέσουμε περαιτέρω ρυθμίσει σε ό,τι αφορά ορισμένα από αυτά τα κρυπτονομίσματα. Ε, τέλος είδαμε κατά πόσο το ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το κατάλληλο για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα, δηλαδή την ε, ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη φοροδιαφυγή, το ξέπλυμα του χρήματος. Και επίσης εξετάσαμε το κατά πόσο έχει νόημα να προσεγγίσουμε γενικότερα σε σχέση με αυτές τις ε, παράνομες δραστηριότητες στην τεχνολογία blockchain. Πώς κάναμε αυτή την εξέταση μέσω desk research. Ουσιαστικά δηλαδή κάναμε έρευνα ε, εγγράφων πολιτικής, νομοθετικά έγγραφα, ε, καθώς και νομικά έγγραφα αλλά και online πηγές σε σχέση με τα κρυπτονομίσματα συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων των ίδιων των κρυπτονομισμάτων και των βασικών παικτών σε αυτό το τομέα. Αυτά από την πλευρά μου και ο, ο καθηγητής ε, Ρούμεν θα σας ε, παρουσιάσει τα πορίσματα. Σας ευχαριστώ. Να σας πω ότι πραγματικά είναι ένας εντυπωσιακό κόσμος αυτός του, του blockchain και των κρυπτονομισμάτων. Ποια είναι τα βασικά μας απορίσματα. Ε, το κυριότερο πόρισμα ή το κύριο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η ανωνυμία. Η ανωνυμία γύρω από τα κρυπτονομίσματα. Και όταν λέω ανωνυμία εννοώ τη ε, συσχέτιση του κάθε χρήστη με την ταυτότητά του. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Η ανωνυμία μπορεί να ε, περιλαμβάνει διαφορετικά είδη ανωνυμίας. Ε, μπορεί να είναι απόλυτη ανωνυμία ή ψευδοανωνυμία. Δηλαδή αν ε, κανείς επενδύσει αρκετή προσπάθεια μπορεί να μάθει ποιος είναι ο χρήστης. Για παράδειγμα το bitcoin είναι έτσι, αλλά άλλα όπως το Monero ή το Dash είναι εντελώς ανώνυμα. Από εκεί και μετά ε, χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο έλεγχος είναι ανεπαρκής με αποτέλεσμα να γίνονται κάποιες ε, μάλλον παράνομες ε, οικονομικές συναλλαγές. Και ε, ακριβώς λόγω της φύσης τους ε, τα κρυπτονομίσματα έχουν εύκολη, δίνουν σε αυτούς τους χρήστες, τους παράνομους ε, χρήστες εύκολη πρόσβαση σε καθαρό χρήμα. Και βέβαια υπάρχει πρόβλημα φόρο γιατί προκειμένου να λάβει χώρα η φορολόγηση μια συναλλαγή, θα πρέπει καταρχήν ο αρμόδιο φορέα να γνωρίζει ότι έχει λάβει χώρα αυτή η συναλλαγή. Και αυτό είναι ακριβώ το πρόβλημα που προκύπτει σε επίπεδο φοροδιαφυγή. Ε, τώρα, το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εντελώς ανεπαρκές ε, σε ό,τι αφορά ακριβώς την, την αντιμετώπιση της ανωνυμίας της χρήσης των κρυπτονομισμάτων. Ε, και εδώ ο συνάδελφος αναφέρθηκε στην πέμπτη αναθεώρηση τη ε, τέταρτης οδηγίας για το ξέπλυμα χρήματο, την οποία θα αναφέρω εγώ με το ακρονίμιο AMLD5. Ε, εκεί λοιπόν γίνεται λόγος για τα εικονικά νομίσματα που κανονικά θα πρέπει να λέγονται κρυπτονομίσματα. Εκεί λοιπόν αναφέρονται συναλλαγές αυτών των ε, υπηρεσιών ή αυτών των νομισμάτων, συγγνώμη, καθώς και υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά την κοινοποίηση ύποπτων συναλλαγών στις αρμόδιες ε, οικονομικές αρχές. Και εδώ βέβαια υπάρχει συζήτηση με, τις, ε, με τη φοροδιαφυγή, γιατί οι εν λόγω πληροφορίε που συλλέγονται για αυτέ τι συναλλαγέ είναι δυνατόν ε, να χρησιμοποιηθούν από τι φορολογικέ αρχέ για να εντοπίσουν φοροδιαφυγή. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα σχετίζονται μεταξύ του, δηλαδή η καταπολέμηση τη τρομοκρατία, η φοροδιαφυγή, το ξέπλυμα χρήματο, όλα του βασίζονται στο να ξεπεραστεί το πρόβλημα τη ανωνυμία. Και μόλι ξεπεραστεί η ανωνυμία μπορούν οι σχετικέ πληροφορίε να διαβιβαστούν στι αρμόδιε κάθε φορά αρχέ. Και από εκεί και μετά απαντήσαμε ε, προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε ένα ακόμα ερώτημα. Ο ορισμός στην πέμπτη αναθεώρηση επαρκεί ε, πάντοτε ο ορισμό των κρυπτονομισμάτων για την αντιμετώπιση ε, τη ε, τρομοκρατία, τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματο. Ευτυχώ θετική ήταν η απάντησή μα. Δηλαδή, ο ορισμό αυτό τη οδηγία επαρκεί. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα κινητό στόχο, αν θέλετε, τα κρυπτονομίσματα. Οπότε θα πρέπει κανεί να εξετάζει τη χρήση τους έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι ο τρέχον ορισμός παραμένει επίκαιρος, παραμένει ικανοποιητικό και καλύπτει επαρκώς τα όσα συμβαίνουν στην αγορά. Περνάω τώρα στο επόμενο κύριο πόρισμά μας. Όταν εξετάσαμε τους ε, κύριους παίκτες εντός εισαγωγικών στις αγορές κρυπτονομισμάτων, διαπιστώσαμε ότι μία σειρά από αυτούς δεν περιλαμβάνονται στην πέμπτη αναθεώρηση της ε, οδηγίας για την καταπολέμηση του ε, ξεπλήματο οικονομικού χρήματο. Πράγμα βέβαια το οποίο αφήνει ορισμένα παραθυράκια, αν θέλετε, στο νόμο σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των σχετικών παρανόμων δραστηριότητων. Ε, και εδώ έχουμε πολλά παραδείγματα, δηλαδή συναλλαγέ ε, μεταξύ κρυπτονομισμάτων, για παράδειγμα, ανταλλάσσει κανεί ένα bitcoin για ένα ether, ε, ή πλατφόρμες έμπορίας των κρυπτονομισμάτων μεταξύ χρηστών και τέτοιου είδους οι πλατφόρμες δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογή, αλλά και άλλοι παροχή ε, πάροχοι υπηρεσιών στο επίπεδο του hardware. Άρα λοιπόν όσοι έχουν δόλια πρόθεση μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα παραστηράκια τη νομοθεσία ε, και να προβούν σε αυτέ τι ε, παράνομες δραστηριότητες με αρνητικά βέβαια αποτελέσματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα διεύνησης του πεδίου εφαρμογή της ε, πέμπτης ε, οδηγία. Και να σα δώσω ένα παράδειγμα. ένα ε, έμπορο ναρκωτικών πουλάει κάποια ναρκωτικά και λαμβάνει χρήματα. Χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα για να αγοράσει μέσω μιας πλατφόρμας τα κρυπτονομίσματα αυτά, τα οποία τα τηρεί σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι το οποίο μόλις αγόρασε και στη συνέχεια προβαίνει σε ανταλλαγή των κρυπτονομισμάτων του, των bitcoins για παράδειγμα, σε ether μέσω μια πλατφόρμα η οποία κάνει ακριβώ αυτό και μόνο, δηλαδή ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων και συνέχεια προβαίνει σε πώληση των ether του μέσω μια ε, πλατφόρμα εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνει και πάλι νομίσματα εναντί αυτών των ether. Όλα λοιπόν αυτά λαμβάνουν χώρα εκτός του πεδίου εφαρμογής της πέμπτης ε, ε, αναθεώρηση τη οδηγία για το εξέβλημα του βρωμικού χρώματο. Άρα λοιπόν όλα αυτά συμβαίνουν στα επέτεινα αν τη νομοθεσία, εκτό δεν καλύπτονται. Τώρα, ένα ακόμα ζήτημα σε ό,τι αφορά την αποκάλυψη της ταυτότητας των χρηστών σε γενικές γραμμές ε, και εδώ αναφέρομαι δηλαδή ε, μόνο σε όσους καλύπτονται από την οδηγία γιατί υπάρχουν για παράδειγμα οι, ε, τα οι, οι αρμόδιοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι ήδη καλύπτονται από τη σχετική υποχρέωση. Αναφέρομαι γενικότερα σε αυτού του ε, παίκτε εδώ και βλέπουμε ότι υπάρχει μία δέσμευση στην πέμπτη αναθεώρηση τη οδηγία ότι η Επιτροπή κατά την επόμενη υπερεθνική αξιολόγηση θα εξετάσει το σύστημα καταχώρηση, η δυνατότητα ενό συστήματο καταχώρηση των χρηστών. Αλλά εμεί φοβόμαστε ότι αυτή η προσέγγιση δεν είναι επαρκή. Εάν δηλαδή ο νομοθέτη θέλει πραγματικά να αποκαλύψει είναι περιγράψει την ανωνυμία των χρηστών των, των νομισμάτων ε, για να ε, καταστήσει την ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας της φοροδιαφυγής και του ξυλούματος σήματος πιο αποτελεσματική, τότε θα πρέπει να αξιοποιηθεί μία από τις δυνατότητες που είχε περιληφθεί στην αξιολόγηση αντικτύπου, δηλαδή η υποχρεωτική εγγραφή και αυτό θέτοντα μια συγκεκριμένη προθεσμία για να το πράξουν. Ε, βέβαια κάτι τέτοιο είναι και πιο παρεμβατικό. Ε, δηλαδή για λόγους ε, αναλογικότητας ε, θα μπορούσε να θέσει κανείς και κάποιες ρήτρε σε ό,τι αφορά την, την, την εφαρμογή, την ουσιαστική εφαρμογή, δηλαδή το σε για ποιον θα πρέπει να ισχύει μια τέτοια υποχρέωση. Γιατί βέβαια δεν μπορούμε να ζητήσουμε να υπάρξει ένα ζήτημα εθελοντική εγγραφή. Δεν μπορούμε δηλαδή να ζητήσουμε από ένα κλέφτη ε, αφού τελέσει αυτή την πράξη να πάει στο αστυνομικό τμήμα εθελοντικά και να δηλώσει ότι προέβη στη διάπραξη ενό εγκλήματο. Άρα λοιπόν όσοι θέλουν να καλύψουν ε, αυτού του ανθρώπου που έχουν αυτέ τι παράνομε δραστηριότητε δεν θα το επιτύχουν μέσω εθελοντικού συστήματο εγγραφή. Ε, τώρα, για κάποια απορίσματα ε, και κάποια ζητήματα πέραν τη εγγραφή των χρηστών θα πρέπει να προβλέψουν ορισμένε απαγορεύσει. Και υπάρχουν εδώ κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχουν δημιουργηθεί δηλαδή για να καταστούσουν ακριβώ του ε, χρήστε ανώνυμου, όπω το Dash, το Μονέρο και άλλα νομίσματα χρησιμοποιούν τεχνολογίε που καθιστούν 100% ανώνυμου του χρήστε του. Ε, και εδώ τίθεται το ερώτημα, πραγματικά χρειάζονται αυτά τα κρυπτονομίσματα ένα τέτοιο βαθμό ανωνυμίας δεν διευκολύνουν υπερβολικά του εγκληματίε. Σε κάθε περίπτωση πάντω η απαγόρευση δεν θα πρέπει να είναι γενικού χαρακτήρα και θα πρέπει αντιθέτω να εστιάζει στα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία δίνουν υπερβολικά, υπερβολικές δυνατότητες ε, στα κρυπτονομίσματα. Τώρα, στο επόμενο σημείο να περάσω. Το ευρωπαϊκό επίπεδο ε, είναι το καταλληλότερο για την μετώπιση των ζητημάτων των κρυπτονομισμάτων, αλλά ακόμα καταλληλότερο το επίπεδο είναι το διεθνέ, βέβαια, γιατί τα κρυπτονομίσματα δεν περιορίζονται από σύνορα ή από περιοχέ. Για παράδειγμα, τα πιο σημαντικά νομίσματα δεν δημιουργούνται, δεν γίνονται mind όπως λέγεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά σε άλλες χώρες, ε, κυρίως στην Κίνα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει διεθνή συνεργασία, ειδικότερα επιβολή κοινών κανόνων σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του ξεπλήματο χρήματο τη τρομοκρατία και ε, τη φοροδιαφυγής και ενδεχομένω και σε επίπεδο G20 θα ήταν πρόσδεκτη μια προσπάθεια. Όπω θα διαπιστώσατε, μέχρι στιγμή αναφέρθηκα μόνο στα κρυπτονομίσματα και όχι στη τεχνολογία blockchain, παρότι αυτό ήταν ο τη παρουσίασή μου, δηλαδή κρυπτονομίσματα και blockchain. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο blockchain. Το blockchain είναι μια τεχνολογία στην οποία βασίζεται η μεγάλη πλειοψηφία των κρυπτονομισμάτων. Αλλά και άλλες εφαρμογές από τον τραπεζικό τομέα. Ουσιαστικά μέσω του blockchain κανείς βγάζει τον διαμεσολαβητή από τη συναλλαγή. Ε, και έτσι δεν χρησιμοποιείται μόνο από τα κρυπτονομίσματα. Και σε κάθε μία περίπτωση το blockchain δεν έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την φοροδιαφυγή, την χρηματοδότηση τη τρομοκρατία ή το ξέπλυμα του χρήματος έχει μία σειρά από χρήσιμες ε, αποχρήσεις ε, στην νόμιμη οικονομία. Άρα λοιπόν οι σχετικέ προσπάθειε για την καταπολέμηση των σχετικών εγκλημάτων δεν θα πρέπει να στραφούν εναντίον του blockchain. Θα πρέπει να στραφούν εναντίον τη παράνομη χρήση τη σχετική τεχνολογία blockchain. Σα ευχαριστώ και αναμένω με ενδιαφέρον ε, τι παρεμβάσει σα ε, και νομίζω πω πρέπει να και 15 δευτερόλεπτα από το χρόνο Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέροντα τα συμπεράσματά σας. Πρέπει προσεκτικά να τα μελετήσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αφετηρία τη μελέτη σας. Και τώρα θα έχουμε δόσεις ερωτήσεων ένα πέντε λεπτά και στη συνέχεια οι απαντήσεις ο συνάδελφος που θέλει να ρωτήσει άπαξ και δεν περνάει το πεντάλεπτο. Ξεκινούμε με τους εισηγητές. Δεν έχουμε τον συνεισηγητή του ΕΛΚΑ, Εγώ είμαι όμως ο άλλος από τους δύο συνεισηγητές. Οπότε θα ξεκινήσουμε την ερώτησή μου και κατόπιν θα προχωρήσουμε ανάλογα με το ποιοι ζητούν το λόγο να καταρτήσουμε μια λίστα με αγορητές. Κύριε Χάουμπεν, μας ε, είπατε, αν κατάλαβα καλά, ότι υπάρχει η στρατηγική των απαγορεύσεων για, χρήση, για κάποιες χρήσεις κρυπτονομισμάτων, ιδίως για τα κρυπτονομισμάτα που συνεπάγονται ανωνυμία. Ε, βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλος παίκτη στην ε, αγορά και μπορεί να καλύψει ε, αυτά τα προβλήματα. Οπότε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς μπορούμε να καλύψουμε, να προωθήσουμε, να υιοθετήσουμε κάποια κρυπτονομίσματα που είναι στα πρότυπά μας. Αλλά βέβαια να ξέρουμε την ταυτότητα των χρηστών τους και θα μας βοηθήσει αυτό σε διάφορες συναλλαγές. Επίσης, αναφέρατε ότι θα πρέπει σε παγκόσμια κλίμακα να γίνει η σχετική ρύθμιση. Και εάν θέλει να δεσπίσει νέους κανόνες για τα κρυπτονίσματα η Ένωση, τότε στο επίπεδο G20 θα υπάρξει κίνητρο, θα υπάρξει όθηση προς τους G20 για να κάνουν και αυτοί κάτι. θα αρχίσω από το τέλος. Ναι, ναι, είπαμε ότι το τέλειο είναι να γίνει παγκόσμια, προσέγγιση παγκόσμια ρύθμιση. Βέβαια, σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία εκκρεμούν Ναι, στο G20 συζητιέται το θέμα. Το FATF επίσης το συζητεί. Άρα το θέμα είναι στα επίκεντρο και επικαιρότητας. Και πρέπει να γίνουν περισσότερα. Θα μπορούσε να γίνει πρωτοπόρα σε αυτή την προσπάθεια νομοθέτησης, δηλαδή η Ένωση. Ήδη βέβαια έχουν γίνει τα πρώτα βήματα. Είχαμε την πέμπτη αναθεώρηση της ε, οδηγίας κατά του ξεπλήματος. Πολύ θετικό αυτό. Όμως λέμε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί η αγορά εξελίσσεται γρήγορα και θα πρέπει με προσοχή να προχωρήσουμε. Γιατί μπορεί αυτά που κάνουμε να είναι ανεπαρκή και ήδη είναι ό,τι έχουμε κάνει ανεπαρκές. Οπότε και αυτοί που θέλουν να παρανομήσουν θα ψάξουν να βρουν τα παραθυράκια. Και υπάρχουν ένα σωρό παραθυράκια στον νόμο. Οπότε εγώ είμαι αναφανδόν υπέρ του να αναλάβει δράση η Ένωση πρωταγωνιστικό ρόλο. Και στη συνέχεια αυτό να επεκταθεί. Αυτά για τη μία ερώτησή σας. Παρακάτω. Ρωτήσατε για το θέμα της απαγόρευσης κάποιων ε, νομισμάτων ή χρήσης νομισμάτων. Είπα για τα πρότυπα της ε, Ένωσης, δηλαδή να έχουμε κριτήριο τη δυνατότητα ανωνυμίας του χρήστη. Αν το πρόβλημα είναι ότι χάνουμε το τρένο τεχνολογικών εξελίσσεων ως ε, νομοθέτες εσείς Έχετε κάποια ιδέα για το πώς θα μπορούσαμε να, να ξεπεράσουμε αυτό μας το πρόβλημα με τι πολιτικές θα μπορούσαμε να προλάβουμε τις εξελίξεις και να μην τρέχουμε από πίσω τους. Να μην νομοθετούμε αργά, κατόπιν ερωτήσεις. Ε, δύσκολο αυτό να σα το απαντήσω, λέει ο κύριο Χάουμπεν. Η δύσκολη είναι ότι όταν κανείς έχει πολλά να κάνει, τότε ε, ρυθμίζει κανεί πράγματα που δεν πρέπει να ρυθμιστούν, οπότε αυτό είναι κακό για το εμπόριο, για την οικονομία. Από την άλλη μεριά, αν κανείς δεν ε, έχει ευρύ φάσμα ρύθμιση, τότε μένουν έξω από τη ρύθμιση εγκληματίε. Άρα, δύσκολη η ισορροπία. Τι να κάνει κανείς για το πρόβλημα. Ε, αυτό είναι το δύσκολο και ίσως κανείς θα έπρεπε να παρακολουθεί τι γίνεται στην πραγματικότητα στην πιάτσα πάρα πολύ προσεκτικά να βλέπει τι παρανομίες γίνονται και να αντιδρά όσο γίνεται ταχύτερα. Ίσως αυτή είναι πιο σωστή προσέγγιση και όχι του να έχει κανείς έναν ευρύτατο ορισμό για το έγκλημα ας πούμε. Όχι, εμείς δεν θεωρούμε ότι η πανάκια είναι η απαγορεύση. Απαγορεύση να υπάρχει όταν το συμφέρον του εγκληματία έχει καταστεί πιο σημαντικό από το συμφέρον της κοινωνίας, της ε, νόμιμης οικονομίας. Να είπαμε αυτή η διαδικασία ανάμειξης για τον τάσο. Ένα κρυπτονόμισμα. Ε, εκεί έχουμε ένα χαρμάνι από διάφορα δεδομένα. Είναι τόσο μπερδεμένα που κανείς δεν μπορεί να διαπιστώσει αν γίνεται χρήση του κρυπτονομίσματος. Πού να βρω λόγους που να δικαιολογούν το ότι αυτό το μπέρδεμα κανείς το χρησιμοποιεί για κάτι άλλο παρά για κάποια παρανομία. Α μου βρει κάποιο. μία εξήγηση νόμιμη χρήση. Εγώ δεν μπορώ. Οπότε η επιβολή απαγόρευση θα πρέπει να είναι καλά στοχευμένη. Όχι, όχι, όχι. Να μην έχουμε ευρύτατε απαγορεύσει. Αλλά και από την άλλη βέβαια, μην δημιουργούμε παραθυράκια για τους εγκληματίες. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά και εσά κύριε Σνάιρ για τα όσα μα ε, είπατε. Και προχωράμε τώρα όσον αφορά τον κατάλογο των ε, εισηγητών. Των, συγγνώμη, τον τον συναδέλφων εδώ που είναι Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σαφές, σαφής η διάγνωση για μένα. Είπατε, το εξηγήσατε ότι τα κρυπτονομίσματα είναι ανώνυμα ε, εξορισμού. Αυτή είναι και η αυτό είναι και το πλεονέκτημα που, έχουν, που προσφέρουν. Επίσης, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται ένα πλαίσιο, μια ευρωπαϊκή νομοθεσία για να παρεμποδιστεί η νομοποίηση παρανομών εσόδων και ότι αυτό ε, συνεπιφέρει. Οργανωμένη εγκληματικότητα, φοροαποφυγή κτλ. Αλλά αυτό που δεν έχω καταλάβει ακόμα καλά είναι το πιστεύετε πραγματικά ότι μπορεί να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο, ένα αριθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να ε, αναιρέσει αυτή τη λογική της ανωνυμίας που χαρακτηρίζει αυτά τα κρυπτονομίσματα και θεωρείται ότι η λογική των κατανεμημένων συστημάτων μπορεί να παρεμποδίσει αυτό το διαβόητο σύστημα της νομοποίησης και ό,τι αυτό συνεπιφέρει. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο, κύριε έχω για να απαντήσετε. Ευχαριστώ για την ε, ερώτηση. Αν πιστεύουμε σε ένα αριθμιστικό πλαίσιο. Ναι. Η απάντηση είναι ναι. Βεβαίω είναι δύσκολο. Ε, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την ανωνυμία. Δηλαδή να αντιμετωπίσουμε κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε. Να πολεμήσουμε κάτι που δεν βλέπουμε και άρα ε, μετατρέπεται σε, μια, σε ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Όταν το βάλουμε σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο πάλι δεν θα μπορούμε να το δούμε. Πάλι στο σκοτάδι θα μένει. Είναι αυτό μειονέκτημα. Ασφαλώς και είναι. Ή μάλλον για να ξαναρχίσω. Όταν θεσπίσουμε μια υποχρεωτική καταχώρηση των χρηστών, τότε ανοίγουμε ένα παραθυράκι στα όσα συμφέρουν, γιατί ο χρήστη πρέπει να είναι καταχωρισμένο. Συμπεριλαμβανομένου και του χρήστη το ε, κρυπτονομίσματος όπως τον τάσκο είναι τελείως ανώνυμο. Μετά όμως περνάω και στη συζήτηση τη σχετική με τη συμμόρφωση και την επιβολή των διατάξεων. Γιατί κάποιος που μπορεί τώρα να είναι κρυφός, μπορεί να θέλει και μετά από μια υποχρεωτική καταχώρηση να μείνει στο σκοτάδι. Πώς θα τον βρούμε αν δεν συμμορφωθεί ο ίδιο με την υποχρέωση καταχώρηση. Ασφαλώς και είναι δύσκολο. Δύσκολο τον βρούμε. Αλλά σημαίνει αυτό ότι ένα αριθμιστικό πλαίσιο είναι άχρηστο. Όχι. Γιατί μας προσφέρεται εργαλεία να αναλάβουμε δράση μόλις το να καλύψουμε αυτό. Αν δεν έχουμε πλαίσιο δεν μπορούμε να δράσουμε. Ενώ αν έχουμε μια εργαλειοθήκη Δηλαδή ενισχύουμε τα εργαλεία που έχουμε στη θέσή μας, την εργαλειοθήκη μας, έτσι ώστε όταν πέσουμε πάνω σε μια παράτυπη χρήση, σε μια αφέμητη μάλλον χρήση, μη νόμιμη χρήση, τότε μπορούμε να αναλάβουμε δράση, πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα. Άρα βεβαίω και χρειάζεται ένα, νομοθετη... ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Δεν θα σώσει την κατάσταση, δεν θα λύσει κάθε πρόβλημα. Αλλά διευκολύνει πολύ γιατί είναι ένα εργαλείο στα χέρια των ε, φορολογικών αρχών, ε, του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αν θα λύσει τα προβλήματα. Καταρχάς, θεωρώ ότι είναι εφικτό ένα σύστημα υποχρεωτική καταχώρησης. Απαγόρευση από την άλλη. Για να περάσω σε αυτό το παράδειγμα. Αυτό είναι δύσκολο. Και μάλιστα πρόκειται και για ευρύτερη δυσκολία, γιατί πολλά από τα νομίσματα αυτά δεν περνούν από μεσολαβητίες. Ε, μόνο μέσω των ε, ε, επικοινωνούν των υπολογιστών κινούνται. Δεν μπορεί κανείς να στοχεύσει έναν υπολογιστή, ή ένα δίκτυο συγκεκριμένο κάπου. Πρέπει να βρούμε κάποιον τον οποίο θα υπαγάγουμε σε μια νομοθεσία και θα είναι αυτό οποίο, κατά το οποίο θα στραφούμε όταν, υπάρχει, όταν υπάρξει μια παράβαση. Όλες αυτές οι τεχνικές βέβαια της ανωνυμοποίησης των ε, νομισμάτων δεν συνδέονται απαραίτητα με ένα φυσικό πρόσωπο ή και νομικό. Αυτό είναι που καθιστά δύσκολη την υπόθεση. Τεχνολογικά είναι μεγάλη πρόκληση. Αλλά πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε να καταστήσουμε παραδείγματι υποχρεωτική την ε, ε, λειτουργία, του, η λειτουργία του συστήματος με έναν διαμεσολαβητή, μεσολαβητή, μια, έναν ενδιάμεσο. Θα μπορούσαμε αυτό, γίνεται, να καταστεί υποχρεωτικό αυτό. Υπάρχουν διάφορε επιλογές που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε. Και με μια επιφύλαξη, αν μου επιτρέπετε, νομική. Απαλλαγή για να δηλώσω ότι δεν είμαι η ε, δήμων στα θέματα τα τεχνικά ω νομικό υποχρεωμένο υποχρεωμένος να κάνω τη διευκρίνηση. Δεν ξέρω ποια είναι η τεχνολογία που θα το εξασφαλίσει αυτό ή πώς θα λειτουργήσει αυτή η τεχνολογία, αλλά είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε σε όρου νομικούς. Κυρία Ρέγνερ, ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ συναρπαστικά όλα αυτά που μας λέτε. Ξέρω βεβαίω. και βλέπω ότι τονίζετε περισσότερο τα νομικά αισθήματα, αλλά θα ήθελα να έρθω σε αυτά που προκύπτουν από την έρευνά σας για να ρωτήσω εάν έχετε καταλήξει σε κάποια στοιχεία ως προς το πέραν της ανωνυμίας που λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί, εάν πέραν της ανωνυμίας είναι χρήσιμα τα, κρυπτονομίσματα. Μπορεί να είναι σε κάτι χρήσιμα. Θα μας δώσετε κάποιες ιδέες. Σε ποιον άλλο στόχο μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλά ωραία και χρήσιμα και πρακτικά ακούμε, αλλά έχετε διαπιστώσει κάτι αυτό. Και κάτι άλλο ως προς το No Air Customer Policy. Ε, υπάρχει κάτι το οποίο διαπιστώνει ότι ήταν ανεπαρκές ως ρύθμιση και χρειάζεται να διευκρινιστεί περισσότερο σε πιο συγκεκριμένους όρους. Παρακαλώ για να απαντήσετε κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ. Αν έχουμε κάνει έρευνα, λέτε, για την αναγκαιότητα του κρυπτονομίσματος. Σας πω, για να είμαι απολύτως ε, πρακτικός και ρεαλιστής, δεν χρειάζεται γιατί έχουμε το ρευστό. Δημιουργήθηκε όμως γιατί οι ε, πολίτες δυσπιστώντας απέναντι στις κεντρικές τράπεζες θέλησαν να φτιάξουν ένα σύστημα δικό τους και ανεξάρτητο από διαμεσολαβητές και κυβερνήσεις. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο εφευρέθηκαν τα κρυπτονομίσματα. Το περίφημο bitcoin νομίζω ήταν η απαρχή, αλλά έχουμε τώρα πολλές εκατοντάδες κρυπτονομισμάτων. Ερώτηση, τα χρειαζόμαστε. Ε, μάλλον όχι, αλλά υπάρχουν. Και καμιά φορά όταν ακούμε τι λέει ο κόσμο που κινείται στην αγορά, όλο αυτό το fintech buzz, ε, γιατί πολλά λέγονται, ε, συχνά ακούμε να λένε ότι α, η μεγάλη καινοτομία δεν είναι τα κρυπτονομίσματα. Μπορεί να είναι φούσκα μόνο. Μπορεί. Η πραγματική όμως καινοτομία και αυτό το ακούω από τους ειδικού του κλάδου, είναι η τεχνολογία, το κατανεμημένο μητρό, οι συστοιχίες, οι πλατφόρμες εθέρα, όλα αυτά είναι πολύ, πολύ σημαντικά η τεχνολογία αυτή, η οποία ουσιαστικά σηματοδοτεί την καινοτομία και από εκεί και πέρα το στοιχείο, το κρύπτο στοιχείο που στηρίζεται πάνω στη τεχνολογία μπορεί να μην το χρειαζόμαστε. Μπορεί και να μην υπάρχει καν σε 10 χρόνια. Ας δούμε. Αλλά όσο υφίσταται τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να το χρησιμοποιήσει ένας εγκληματία. Αυτό είναι δεδομένο ότι υπάρχει. Και είναι δεδομένο επίσης ότι μπορεί να χρησιμοποιείται ή ήδη χρησιμοποιείται από εγκληματίε. Αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Στο δεύτερο ερώτημα, αν καταλαβαίνω καλά, συνοψίζοντας, ρωτάτε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε το ισχύον πλαίσιο. Το ισχύον πλαίσιο έχει ως εξή. Έχουμε την ε, επερχόμενη οδηγία για την καταπολέμηση παρανομών εσόδων, την 5, την AMLD, ε, που δεν έχει ακόμα αρχίσει να εφαρμόζεται γιατί ισχύει ακόμα η 4, η 5. Αυτή τη στιγμή πέραν αυτού δεν έχουμε τίποτα, δεν καλύπτει δηλαδή τίποτα έχουμε την οδηγία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά πληροφορίε μπορούν να τα αλλάξουν οι, οι αρχέ μεταξύ του μόνο αν τι έχουν στα χέρια του. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν πληροφορίε τέτοιου τύπου, γιατί είναι ανώνυμα όλα αυτά τα στοιχεία. Επομένω, δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μα. Άρα μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση και ήδη βελτιώνεται από την ε, πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση, γιατί σε αυτήν περιλαμβάνονται τα εικονικά ε, νομίσματα και οι ανταλλαγή και οι ε, custodian providers, αυτοί δηλαδή οι οποίοι παρέχουν την δυνατότητα των συναλλαγών παρακολουθώντας την πορεία του νομίσματος. Άρα λοιπόν με αυτά τα δύο στοιχεία ήδη έχουμε ρίξει αρκετό φως γιατί είναι, ε, έχουμε το στοιχείο της ε, υποχρέωσης δέουσας επιμέλειας. Και άρα είναι υποχρεωμένη η αρχή που θα εντοπίσει κάτι να ε, διοχετεύσει τις πληροφορίες και να τις φτάσει μέχρι η φορολογική αρχή, εάν χρειάζεται ε, μπορεί να βελτιωθεί το σύστημα. Ασφαλώς και αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματά μας. Υπάρχουν παράγοντες στην αγορά που δεν καλύπτονται από αυτήν την νομοθεσία και προσπάθησα να το εξηγήσω αυτό με ένα παράδειγμα ότι εάν ε, χρησιμοποιώ μια ε, πλατφόρμα τύπου ανταλλαγή peer-to-peer από μεταξύ ισοτήμων, δηλαδή ε, μια ε, ιστοσελίδα, ένα ιστότοπο μεταξύ, που συνδέει τους χρήστες μεταξύ τους. Να πω, πω πάω σε ένα μπαρ στι Βρυξέλλες και θέλω να αγοράσω bitcoin. Αυτό μπορώ να το κάνω μέσα από, μια, από ένα συναλλακτήριο ηλεκτρονικό. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτή η πλατφόρμα, η συναλλακτική δεν καλύπτεται. Η καθαρή κρυπτο κρυπτογραφημένη ε, πλατφόρμα πάλι δεν καλύπτεται. Εάν δηλαδή έχει κάποιο Stellar, Bitcoin, Ether, οποιοδήποτε άλλο, α πιάσουμε την ονοματολογία των 10 κρυπτονομισμάτων με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση τη αγορά. Οποιοδήποτε από αυτά τα νομίσματα λοιπόν να θέλω να ανταλλάξω για να πάρω ένα άλλο κρυπτονόμισμα, μπορεί να συμβεί αυτό. Και να συμβεί εκτός του ρυθμιστικού πλαισίου. Γιατί αυτές οι συναλλαγές δεν καλύπτονται από την πέμπτη οδηγία. Και μάλιστα κάποιοι λένε ότι θα πρέπει στο miner, στον εξορίκτη, όχι τον πελάτη δηλαδή, να επιβληθεί αυτή η, υποχρέωση. Mining τι σημαίνει. Σημαίνει ότι παράγω με την δύναμη την υπολογιστική των κομπιούτερ μου, των υπολογιστών μου, όπως βλέπουμε με τα μεγάλα συστήματα, που τα μεγάλα δίκτυα μάλλον στην Κίνα, παράγω bitcoin, η κρυπτονόμισμα. Αν λοιπόν μπορεί κάποιος να πουλήσει αυτά τα νομίσματα ως miner, τώρα το πάλι ξεφεύγει από τον έλεγχο, πάλι μένει στο σκοτάδι στη σκοτεινή πλευρά. Επομένως, υπάρχει μια σειρά από κρυπτονομίσματα που δεν καλύπτει ακόμη η ευρωπαϊκή νομοθεσία και υπάρχει μεγάλο περιθώριο να αξιοποιήσει ένας ε, εφάνταστος εγκληματίας και να μείνει πάλι ε, στο σκοτάδι. Ευχαριστώ. Η, CR η σειρά της CR τώρα, αλλά δεν ξέρω αν εκπροσωπείται από κάποιον. Ο Βόλφαν κλείνει λοιπόν για τους ε, φιλελεύθερους. Ε, σας ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι ε, σοκαρίστηκα όταν μας είπατε πως οι ζημίες από τη χρήση των κρυπτονομισμάτων ανέρχονται σε 7 δισεκατομμύρια. Δηλαδή ήξερα ότι είναι μεγάλη ζημία, αλλά πραγματικά το να υπερβαίνει τα 7 δισεκατομμύρια είναι εξοργιστικό και θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Όποτε υπάρχει μια τεχνολογική καινοτομία, είναι πολύ δύσκολο να τη σταματήσει κανεί. Όταν προσπαθεί καλή να κάνει κάτι τέτοιο, θα συνεχίσει να αυξάνεται. Οπότε το ερώτημα που τίθεται είναι τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ θυμάμαι πως αυτό που διαβάζω κατά τους τελευταίους 6, 8, 9 μήνες ήταν ότι πολλές τράπεζες εξέτασαν το ενδεχόμενο του να απαγορεύσουν τα κρυπτονομίσματα και εσείς ε, έμεσα απαντήσατε στο ερώτημα που ήθελα να σας θέσω ότι δεν θεωρείτε πως κάτι τέτοιο είναι δυνατό γιατί ακριβώς τα κρυπτονομίσματα είναι ανώνυμα. Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι πραγματικά αδύνατο κάτι τέτοιο. Οπότε το ερώτημα που θέτω είναι αντί να σκεφτόμαστε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα θετικό πλαίσιο, μήπω θα πρέπει να πούμε ότι είναι παράνομη χρήση των κρυπτονομισμάτων. Δηλαδή ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιείται για παράνομε δραστηριότητε το κρυπτονόμισμα, ενδεχομένω θα μπορούσαμε να απαγορεύσουμε πλήρω τη χρήση του. Είναι και αυτή δηλαδή μια δυνατότητα, ειδικότερα αφού οι μεγάλε τράπεζε εξέταζαν αυτό το ενδεχόμενο τη πλήρου απαγόρευση. Από ό,τι ξέρω, πάντω δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Από εκεί και μετά υπάρχει μια περαιτέρω πτυχή δεν είναι δηλαδή μόνο η οικονομική ζημία που οποία η χώρα με τη χρήση των κρυπτονομισμάτων, αλλά ταυτόχρονα υπονομεύεται η εμπιστοσύνη στο χρηματοοικονομικό σύστημα που έχουμε και ειδικότερα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ε, χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό σύστημα και αν επιτρέψουμε στα κρυπτονομίσματα να καταστρέψουν την εμπιστοσύνη των πολιτών μας σε αυτό το σύστημα ε, τότε αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για την κοινωνία μας γιατί τελικά μπορεί να τα καταφέρουν μπορεί δηλαδή να διαβρωθεί η εμπιστοσύνη ξεκινώντας από ένα από μια μικρή ομάδα ατόμων που λένε ότι δεν πιστεύουμε στην, στο μεγάλο τραπεζικό, το κεντρικό τραπεζικό σύστημα, δημιουργούμε τη δική μας τεχνολογία και ούτω καθεξής, μπορεί αυτό το σκεπτικό να εξαπλωθεί και κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ένα τεράστιο κίνδυνο για την κοινωνία και βέβαια αυτό θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που θα αναθέσω. Τώρα το δεύτερο. Ε, οι διακυμάνσεις που, ε, τις οποίες υφίσταται ένα ε, κρυπτονόμισμα είναι τεράστιες. Δηλαδή μπορούν να πάνε από 20.000 σε 10.000 και οτιδήποτε άλλο. Οπότε πραγματικά είναι τεράστιες αυτές οι διακυμάνσεις. Μήπως λοιπόν θα ήταν δυνατό να αξιοποιήσουμε το σύστημα έτσι ώστε εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα να πλήττονται πραγματικά από τον ε, κίνδυνο αν αυτός ε, προκύψει. Δηλαδή, ε, όσοι χρησιμοποιούν τέτοιο είδο νομίσματα, όταν αυτά χάνουν σε αξία, να νιώθουν πολύ έντονο αυτό το αρνητικό αντίκτυπο, έτσι ώστε να αποθαρρύνονται από τη χρήση του. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο, ο κύριο Ρουβέν έχει και πάλι το λόγο. Σα ευχαριστώ και αντιλαμβάνομαι πλήρω το σκεπτικό σα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την απαγόρευση των κρυπτονομισμάτων και το αν είναι τελικά αδύνατη ή όχι, νομίζω πως δεν είναι αδύνατη. Γιατί αυτό που έχει καταδείξει η δική μας ταξινομία είναι ότι δεν είναι όλα ίδια τα κρυπτονομίσματα. Δηλαδή, ορισμένα μπορούν να απαγορευτούν εύκολα, γιατί μπορούν να αναγνωριστούν ακριβώ και μπορεί κανεί να επιβάλλει την απαγόρευσή του, αλλά υπάρχουν άλλα όπου δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει αυτό. Υπάρχουν εκατοντάδες διαφορετικών κρυπτονομισμάτων και το κάθε ένα από αυτά με τα δικά του χαρακτηριστικά. Οπότε η απαγόρευση εξαρτάται από τη φύση, από την ιδιαιτερότητα αν θέλετε του κάθε κρυπτονομίσματος. Κάποια λοιπόν είναι ευκολότερο και κάποια δυσκολότερο να απαγορευτούν. Τώρα αυτό που είπατε ότι ορισμένε τράπεζε εξέτασαν το ενδεχόμενο απαγόρευση των κρυπτονομισμάτων. Έχω προετοιμάσει μια, είχα μάλλον διαβάσει μια μελέτη το 2015 από Ευρωπαϊκή ε, και η παγκόσμια ε, οπτική γωνία και ήρθα σε ε, επαφή με τις τραπεζικές αρχές του Βελγίου, οπότε εξέτασα το ζήτημα και από τη δική τους οπτική γωνία, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, αλλά οι τράπεζες δεν είπαν ότι θέλουν να γίνει μια απαγόρευση, απλώς ήταν πάρα πολύ επιφυλακτικές απέναντι στην τοποθέτησή τους. Δηλαδή δεν τοποθετούνται δημοσίες γιατί θέλουν να δουν πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντω η απαγόρευση παραμένει μέσα στι δυνατότητε. Το αντίθετο ωστόσο επιχείρημα, δηλαδή κατά τη απαγόρευσης, είναι ότι και τα χαρτονομίσματα, δηλαδή τα ρευστά, είναι εντελώ ε, ανώνυμα. Εντελώς ανώνυμα είναι. Άρα λοιπόν τι θα πρέπει να κάνουμε, να απαγορεύσουμε και το ρευστό. Αυτό ε, που μπορούμε να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε την νομοθεσία που υπάρχει σε ό,τι αφορά το ξέπλυμα βρωμικού χρήματο. Δηλαδή πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο χρημάτων, πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό, εάν κανείς διαβαίνει με αυτό το ποσό τα σύνορα θα πρέπει να το δηλώνει. Άρα λοιπόν, δεν χρειάζεται να επιβληθεί μια απαγόρευση, αλλά θα πρέπει κανείς να ελέγξει το τι συμβαίνει. Έτσι ώστε να μπορεί να στοχεύει ακριβώς σε αυτές τις περιπτώσεις παράνομης χρήσης. Μετά, σε ό,τι αφορά τις διακυμάνσεις του νομίσματος. Εδώ ερχόμαστε στον τομέα της ε, νομοθεσία ό,τι αφορά τις χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίες. Τη σήμερα ημέρα τα πράγματα ε, έτσι όπως έχουν θα πρέπει να δει κανείς την ε, σχετική νομοθεσία για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τα securities και να εξετάσει καταρχήν αυτό το οποίο, με το οποίο ασχολούμαι εδώ είναι security ή όχι. Ε, αλλά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ω τέτοιο. Και από εκεί και μετά, για τα προσπέκτου, για παράδειγμα, η οδηγία χρειάζεται να υπάρχει ένα εκδότη, αλλά δεν εκδίδει κανεί το κρυπτονόμισμα. Μετά, σε ό,τι αφορά την ε, την οδηγία, σε ό,τι αφορά τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Ε, και πάλι εδώ δεν έχουμε μια καταχωρημένη επιχείρηση ω πάροχο αυτών των υπηρεσιών. Οπότε υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο, αλλά ε, για να είμαι απολύτω ειλικρινή μαζί σα, τα κρυπτονομίσματα καταφέρουν να μην υπάγονται σε καμία από αυτέ τι νομοθεσίε που υπάρχουν. Και γι' αυτό η EBA προτείνει μία πιο ευρία προσέγγιση και προτείνει αυτή η επέκταση των εισαγωγικών των κρυπτονομισμάτων να δημιουργήσουν ήδη ένα σύστημα αδειοδότησης το οποίο με την παράδοση του χρόνου θα μπορούσε να αποτελέσει μια, μια καλή εναλλακτική. Γιατί βέβαια θα κάλυπτε και περαιτέρω ζητήματα ε, πέραν του ξεπλήματος ε, βρώμικου χρήματος. Αν δηλαδή θέλει κανείς να συμπεριλάβει πέρα από το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος και τη φοροδιαφυγή, θέλει να περιλάβει και την προστασία των επενδυτών, τότε θα πρέπει να ε, προσθέσει ακριβώς και σύστημα εγκρίσεων με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τους διευθυντές και τους μετόχους ελάχιστες κεφαλαίες απαιτήσει και ούτω καθεξής. Αυτά σε ό,τι φορά τις ανησυχίες που εκφράσατε. Ευχαριστούμε πολύ καθηγητά. Προχωρούμε τώρα. Η Ντανούτα Γεσλοδιέτσκα έχει σειρά σύμφωνα με τη λίστα. Όχι, όχι, όχι, όχι για τώρα. Θα ήθελα να μιλήσω μετά. Ε, Τώρα για το ΚΑΤΣΔΙΑΕ, η Νίνα Γκίλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ήξερα ότι είμαι στη λίστα του ΚΑΤΣΔΙΑΕ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Σας ευχαριστούμε για τις εισήγησει σας και νομίζω ότι μας εξηγήσατε τις ευκαιρίε, τα προβλήματα και νομίζω ότι πρόκειται για κάτι καινούριο στο οποίο έχουν στρέψει την προσοχή τους οι διοίκες, οι νομοθέτες κλπ. Και βλέπουμε Γαλλία και Γερμανία ήδη έχουν λάβει συγκεκριμένα μέτρα. Και νομίζω όμως ότι θα πρέπει να προσέξουν περισσότερο το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλό σκοπό η τεχνολογία. Να, ε, παράδειγμα, η εφορία μπορεί να έχει κάποια ευφύ εφαρμογή ούτω ώστε να <clears throat> αυτό το, αυτή η υπηρεσία και το εργαστήριο ξέρω εγώ να χρησιμοποιήσει το υπολογιστικό νέφος και διάφορα άλλα ε, για αιτήσει, για, για αποστολή ειδοποιήσεων της εφορίας και εντάξει Καλά μας τα είπατε. Θέλουμε να καταπονήσουμε την απάτη. Από την άλλη μεριά όμως να μην φημώσουμε, να μην κόψουμε το δρόμο στην καινοτομία. Να, να δούμε τι έχει γίνει, τι έχει θεσπιστεί όπως αυτά που γίνανε στην ε, Μάλτα. Τι να κάνουμε. Να, κατα... να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα των Κινέζων για την πολέμηση της ε, φοροδιαφυγής. Πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Επίσης κάτι άλλο για το blockchain. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά τα δεδομένα. Αλλά τι γίνεται με το GDPR. Πώς μπορούμε αυτό να το συντεριάξουν το GDPR. Ας πούμε. Ένα σωρό ερωτήσει ε, καθηγητά. Χάουντεν, ναι, ναι, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μόνο που είναι εκτός θέματος κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν τα περιείχε η μελέτη μας, τέλος πάντων. Πάντως ε, θα τα μελετήσω και θα σας πω. Θα σας στείλω την απάντηση μου γράφω τώρα. Ήθελα να πω ότι σίγουρα είμαστε στο δύο κύματο για την χρήση της τεχνολογίας. Η τεχνολογία θα πρέπει να αφαιθεί, να προχωρήσει. Ε, απλώς θα πει κανεί κάτι να κάνει για την παρανομία. Άρα, πόλεμος όχι στην τεχνολογία, αλλά στην παρανομία. και το blockchain θα μπορούσε να ε, αντικαταστήσει τα παραδοσιακά μητρώα όπου, να, πώς έκανε το Delaware να πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα η οικονομία άρα ας μην πανεύουμε και ας αφήσουμε την τεχνολογία να επιβιώσει, να προχωρήσει για να καταπολεμήσουμε επομένω το έγκλημα και όπως σας είπα είναι ένα θαυμαστό κόσμος ε, και ρίχνοντα κανεί μια ματιά σε κάποια από αυτά τα νομίσματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει πώ λειτουργούν ποια είναι τα χαρακτηριστικά του τα βασικά οπότε είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς το ίδιο το νόμισμα από την τεχνολογία να τα ξέρει εδώ καλύτερα ο Αλεξάνδρ το Ethereum, το Ethereum είναι μια τεχνολογία, είναι μια πλατφόρμα, πλατφόρμα για εφής συμβάσεις. Αλλά υπάρχει και ένα κρυπτονόμισμα που την υποστηρίζει την πλατφόρμα, μάλλον την, την, την τροφοδοτεί, που είναι το Ether. Αλλά το Ethereum, η πλατφόρμα, μπορεί να είναι αντικείμενο εμπορίας χωριστά. Επομένως είναι και τεχνολογία και κατά κάποιο τρόπο νόμισμα. Ε, για αυτό ε, ξεπηδάνε όλες αυτές οι δυσκολίες. Τι να σας πω, δεν είναι και τόσο εύκολο να σας απαντήσω πιο απλά πάντα. Ε, οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε κάθε κράτος. Έχουμε ήδη πάνω από 90 σελίδες μελέτη. Πάντως εμείς δουλέψαμε στη βάση του τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα το τι γίνεται στην Κίνα. Δεν τα ξέρω τόσο καλά εκείνα τα θέματα αλλά ξέρω ότι είτε πρόκειται να απαγορεύσουν είτε ήδη έχουν απαγορεύσει τα κρυπτονομίσματα. Τώρα τη σχέση αυτών με το GDPR και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Ε, ο κύριος Σέιβερς. Από ό,τι ξέρω έχουμε την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών και το 17 δημοσιοποίησε κάποια έκθεση για κρυπτονομίσματα τα οποία τα, τα κόβει, τα δημιουργεί κάποια κεντρική τράπεζα. Άρα θέλουν να δούνε τι γίνεται με την τεχνολογία του blockchain και εκείνη. Πώς θα μπορούσε να υπάρξει αξιοποίηση σε ευρύτερη κλίμακα. Να, τι αξίζει να ερευνηθεί. Σας ευχαριστώ και τους δύο, Πρόεδρος, και σας ρώτησε πολλά η Νίνα Γκίλ και αν νομίζετε ότι μπορείτε απαντήστε τις εγγράφως. Γιατί ακόμα και αν είναι εκτός ε, μελέτης σας ε, αξίζουν αυτές οι ερωτήσεις. Προχωρούμε τώρα. Για το έλεγχο, ο κύριος Διντιέ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για να επανέλθω στη συζήτηση που είχαμε τώρα και τη δυνατότητα να απαγορέψουμε ή όχι τα κρυπτονομίσματα. Καταρχάς μου φαίνεται ουτοπικό. Και δευτερευόντως, δεν ξέρω καν αν είναι επιθυμητό, ε, διότι ε, εάν το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, δεν σημαίνει πρέπει να καταργήσουμε το σύστημα. Πρέπει να το ρυθμίσουμε. Και αυτή είναι και η αποστολή μα. Ε, από την άλλη, αντιλαμβάνομαι και ποια είναι η δυσκολία του εγχειρήματο, και εδώ απευθύνομαι όχι μόνο στου καθηγητέ αλλά και του συναδέλφου. Η δυσκολία λοιπόν του εγχειρήματο, διότι πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο δύσκολα ελέγχεται περιγράφεται, συγκρατείται, γιατί είναι αόριστο, γιατί είναι διάχυτο, αόρατο και το πώς θα ρυθμίσουμε το αόρατο ή πώς θα υλοποιήσουμε τη ρύθμιση του αόρατου αγγίζει τα όρια του ανέφικτου. Κυρία καθηγητά, αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθείτε τουλάχιστον να περιγράψετε κάτι το περίπλοκο. Από την άλλη, πριν από λίγο αναφερθήκατε σε ενδιάμεσους Υπάρχει ο Γενικός ε, Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων. Με τον ε, Data Protection Officer, DPO, τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που σε κάθε επιχείρηση είναι αρμόδιος για την ε, επιβολή, την εφαρμογή αυτής της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος ώστε να εγκαθιδρυθεί ένας διαμεσολαβητής, σε διάμεσος καλύτερα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μέσα σε αυτή την ιδέα του αόρατου, του άειλου, του ανώνυμου, δηλαδή του κρυπτονομίσματος, για να προσωποποιήσουμε κάπως και να εξορθολογήσουμε αυτό το σύστημα. Μπορεί να σας φαίνεται αφελές το ερώτημα, αλλά προσπαθώ να, αντιληφθώ σε ποιο βαθμό είναι δυνατόν αυτό και εφικτό. Ο πρόεδρος ευχαριστώ πολύ, ο καθηγητής κύριος Χόμπεν. Ευχαριστώ πολύ για την ε, συμπληρωματική ερώτηση. Συμφωνώ απολύτως ότι δεν πρέπει να απαγορεύσουμε ή να καταστρέψουμε κάτι, αλλά να το ρυθμίσουμε. Ε, αν ε, πρόκειται για απαγόρευση, θα πρέπει να είναι πολύ περιορισμένη και ειδική. Αν πρόκειται για απαγόρευση των κρυπτονομισμάτων, αυτή, αν επιλεγεί δηλαδή η απαγόρευση των κρυπτονομισμάτων, αυτή θα αφορά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτά δηλαδή τα οποία επιτρέπουν χωρί κάποια άλλη ε, στόχευση ή χρησιμότητα, υπερβολικό περιθώριο κινήσεων στους εγκληματίες. Αλλά κατά τα άλλα δεν χρειάζεται παρά μόνο μια γενική πλαισίωση και ρύθμιση, όχι απαγόρευση, πράγμα το οποίο ούτως ή άλλως μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίζει με τη Γενική Οδηγία για την Καταπολέμηση Παράνομων Εσόδων, αλλά πάλι που χρειάζεται μια συμπλήρωση, όπως άλλωστε μας λέει και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Για τον Μεσολαβητή. Όχι, δεν είναι αφελής καθόλου η παρατηρήσή σας. Τουραντίον μάλιστα. Πρόκειται για μια από τις επιλογές που μπορούμε να εξετάσουμε. Αν δεν υπάρχει πρόσωπο στο οποίο να μπορούμε να στραφούμε, ας το δημιουργήσουμε. Να μην μπορεί κανείς να αναλάβει δραστηριότητα την ε, αγορά αυτή, εάν δεν υπάρχει πρόσωπο με το οποίο να μπορεί να επικοινωνήσει κανείς. Και αν δεν υπάρχει ο απεύθυνο να κλείνει ε, το κομμάτι αυτό της αγοράς. Αυτή μπορεί να είναι η λύση για τα νομίσματα αυτά, τα οποία ξεπερνούν κάθε εξορθολογισμό, όπως λέτε κι εσείς. Και βεβαίως είναι όλες αυτές οι πτυχές. Τα και βλέπετε ότι κάποια από αυτά είναι ψηφιακά. Καταρχήν δεν υπάρχει κάποιος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στο, στο, στον υπολογιστή και κάποια άλλο όπως το καρντάν υπάρχουν κάποιοι που κινούν τα νήματα οι οποίοι είναι δυνατόν να ε, κάτω ονομαστούν να επισημανθούν και υπάρχουν κάποιοι φορεί πίσω από αυτά τα νομίσματα που τα φτιάχνουν οπότε εκεί είναι πιο εύκολο όμως ε, βέβαια δεν είναι εκεί το πρόβλημα δεν γίνεται εκεί η παρανομία άλλα είναι αυτά που είναι πιο φευγαλαία οπότε αυτά θα πρέπει να διευκολύνει να συγγνώμη διερευνήσει κανείς και το να υπάρχει ενδιάμεσο αυτό είναι μια καλή λύση. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Κόφοδ. Α, αυτό καλύπτει και αυτό που έλεγα εγώ για τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο κύριο Τόρβαλ. Σα ευχαριστώ. Ε, βέβαια και τα έχουμε μπερδέψει. Και εμείς και εμείς όλοι δυσκολευόμαστε γιατί πριν από λίγες μέρες υπήρχε τίτλος στους Financial Times και έλεγε για το πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει γίνει, το πώς κανείς μπορεί να διερευνήσει εδώ τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, αλλά θα μπορούσαμε να δανειστούμε κάποιε παλιότερε έννοιες για να βοηθηθούμε, είπατε, σε κάποια φάση σκεφτείτε ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στη, στην πιάτσα. Όμω, δεν υπάρχει πιάτσα. Πού να την βρούμε δεν υπάρχει κάποιος χώρος με αυτή την έννοια την παλιά. Είναι το νέφος, το cloud. Και πώς θα δώσει κανείς τον ορισμό σε αυτή την περίπτωση του cloud. Όμως, για να πούμε που υπάρχει δικαιοδοσία, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος χώρος για να ασκηθεί αυτή Άρα έχουν άλλη έννοια. Μάλλον είναι διαφορετικέ. οι, δεν είναι παραδοσιακέ οι έννοιε που ισχύουν. Και το δικαιοδοσία λοιπόν έχει άλλη έννοια προκειμένου. Πάντως ευχαριστούμε για όσα είπατε. Ε, κύριε καθηγητά, κύριε Χάουντερ, ε, βέβαια και συμφωνώ μαζί σας ότι είναι δύσκολο να παρακολουθήσει κανεί πώ εξελίσσονται όλα αυτά, γιατί δεν πρόκειται για τον υλικό χειροπιαστό κόσμο Ω επιτοπλιστών. Όμως θα να κάνουμε κάτι για να καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί αυτά γίνονται και ε, γίνονται και με παράνομο τρόπο πολλές φορές. Οπότε φυσικά και είναι αυτά πολλές φορές εκτός της φυσιολογικής ένομης τάξης, αλλά ακριβώς μια που δεν είναι κάτι χειροπιαστό ε, γίνεται πιο δύσκολο. Αλλά δεν είμαι τεχνικός, τεχνοκράτης, τέλος πάντων, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, αυτοί κάτι θα μπορούσαν να σκαρφίσουν και να βρουν ένα παράδειγμα από το bitcoin το οποίο το προωθούσαν ως ανώνυμο. Και μετά από το MIT κάποιοι ερευνητέ τα κατάφεραν. Κάπως τα κατάφεραν πάνω στην πλατφόρμα blockchain να συνδέσουν την χρήση του bitcoin σε κάποιον που θα μπορούσε να ταυτοποιηθεί, να επισημανθεί. Επομένως, πάει η πλήρης ανωνυμία. Μπορούμε τώρα να βρούμε έστω και δύσκολα ε, την ταυτότητα του χρηστή. Εντάξει, είναι δύσκολο, περίπλοκο, χρειάζεται know-how. Οπότε, για να προχωρήσει κανείς, είναι δύσκολο. Πάντως, αισιοδοξία ότι είναι εφικτό αυτό. Όχι, δεν θα το κάνω εγώ αυτό, κάποιος άλλος, αλλά υπάρχουν η δίκη προς το κύριο Θόρβολτς εκτός ε, μικροφώνου. Α, αυτό που είπατε για το ότι κάθε ένωμη τάξη χρειάζεται έναν ε, χώρο. Όχι, τα κρυπτονομίσματα δεν περιορίζονται από σύνορα, από όρια. Βέβαια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ευρωπαϊκός χώρος είναι κατάλληλος, καλύτερος από τον εθνικό, αλλά Πρόκειται για το παγκόσμιο, το διεθνές επίπεδο, για ό,τι κάνουμε. Αυτό είναι το άριστο. Άρα αυτό και είναι το πιο δόκιμο, το πιο αποτελεσματικό. Κάτι να γίνει σε διεθνές επίπεδο. Ε, ευχαριστούμε καθηγητά, λέει ο Πρόεδρος. Τελευταία ερώτηση για αυτή τη φάση. Λουμίσελ. Ναι, μια πρώτη ερώτηση καταρχάς. Πώς συνεργάζεται με τη Europol και την Interpol η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, θέσει ένα τέρμα ε, στον ηλεκτρονικό εκβιασμό και τα λίτρα που ζητούνται και που πληρώνονται με μέσον το bitcoin. Επίσης, μήπως θα ήταν πιο ασφαλές να ε, φτιάξουμε εικονικό νόμισμα, επίσημο θα το πω έτσι, ώστε να τεθεί υπό τον έλεγχο μιας κεντρικής τράπεζας και να είναι πιο ασφα... και πιο ασφαλές. Επίσης, το Τιτάνιο ως έργο που έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με 5 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση που στόχο έχει να θέσει τέρμα σε ε, πρακτικές ε, ύποπτες, χρηματοδότηση τρομοκρατίας, ε, ξέπνιμα χρήματος κλπ. Πού βρίσκεται, Απλέ ερωτήσεις, συγκεκριμένε περιμένω απαντήσει. Ευχαριστώ και τελευταίο γύρος, κύριε Χόβπεν. Ναι, όντω ε, πολύ συγκεκριμένε ερωτήσεις, αλλά δύσκολε. Επιτρέψτε μου στις δύο να δώσω γραπτές απαντήσεις στη χρήση του blockchain ε, για τη χρήση ηλεκτρονικών λίτρων και το titanium για την ε, δημιουργία νομίσματος από κεντρική τράπεζα κρατικού δηλαδή, ασφαλώ αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση ώστε να ξεφύγει και από το σκοτάδι. Αυτό δηλαδή είναι μια λύση που θα μπορούσε να διερευνηθεί, αλλά αλλά αυτό θα γινόταν σε παραγνώριση του λόγου για τον οποίο δημιουργήθηκε το κρυπτονόμισμα. Και αυτή, αυτός ο λόγος, αυτή η λόγη ήταν ότι ο κόσμος δεν εμπιστευόταν την κρατική εποπτεία και την διαχείριση των νομισμάτων από τις κεντρικές τράπεζες. Άρα ναι, υπάρχει δυνατότητα. Ρυθμιστικά να επιβληθεί αυτό. Αλλά αντίκειται σε όλη τη λογική και τη φιλοσοφία του κρυπτονομίσματος. Και ίσως αυτό να έχει σε συνέπεια ότι μπορεί και να το καταστρέψει. Μπράβο, επιτρέψτε μου όμως να τα ξανασκεφτώ και να επανέλθω γραπτός. Καλώς ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, ε, κύριε καθηγητά, κύριε Σάιας, για τη μελέτη σας και τις απαντήσεις σας. Και βέβαια για την υπόσχεση να μας δώσετε και γραπτές απαντήσεις. Θα τις περιμένουμε. Τώρα λοιπόν μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο πάνελ μας. σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στα διεθνή φορολογικά ζητήματα, τις προκλήσεις ε, και τα ε, και τους τρόπους τους, ε, έχουμε δύο ομιλητές εδώ, την κυρία Έλλη Χατζίεβα που είναι η ιδρύτρια και διευθύντρια του Dialogue for Europe, Διάλογος για την Ευρώπη. Έχετε το λόγο λοιπόν. Πρόεδρε, συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Οι προηγούμενες συνάδελφοι, οι προηγούμενοι ομιλητές αναφέρθηκαν στα κυριότερα ζητήματα σε σχέση με την οικονομία, ε, τα οποία βέβαια ταυτόχρονα θέτουν πολύ σημαντικά φορολογικά ζητήματα. Η ψηφιακή οικονομία αυξάνεται με δραματικούς ρυθμούς και επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας. Ε, τα ψηφιακά αγαθά βέβαια είναι εξαιρετικά ε, κινητά και κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να έχουν φυσική παρουσία στην χώρα στην οποία γίνεται η εμπορία τους. Εδώ υπάρχει μεγάλος αριθμός αγαθών με περιεχόμενο που δημιουργείται από τους ε, χρήστες. Οπότε, εγώ στη δική μου ε, προηγούμενη μελέτη προσπάθησα να θέσω μια κατηγορία σε αυτό το είδος τα ψηφιακά αγαθά, αλλά τώρα μετά από δύο χρόνια πρέπει να αναθεωρήσω αυτή την κατηγοριοποίηση, γιατί μεγάλοι ε, πάροχοι, όπως για παράδειγμα η Amazon, έχουν μια σειρά από διαφορετικά αγαθά και διαφορετικά είδη επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται. Ε, για παράδειγμα το Netflix ε, ήταν ε, καταρχήν μόνο μεταπολιτής ενώ τώρα το ίδιο το Netflix προβαίνει στην παραγωγή ταινιών και μετά βλέπουμε ότι μια σειρά από περαιτέρω κλάδι ψηφιοποιούνται και αυτοματοποιούνται λένε και περισσότερο όπως για παράδειγμα η αυτόματη οδήγηση. Άρα λοιπόν εδώ μας ενδιαφέρει πολύ η φάση της, το ζήτημα της δημιουργίας της αξίας και της αλυσίδα της δημιουργίας αξίας. Είναι δύσκολο λοιπόν να καθαρίσουμε το ε, τι ακριβώ είναι αυτό τα ψηφιακά αγαθά που δημιουργεί την αξία. Κάποια έχουν ονομάσει τα ψηφιακά αγαθά ω το πετρέλαιο τη δική μα εποχή. Αλλά είναι πραγματικά δυνατό να, να πούμε πού ακριβώς δημιουργούν και πώς, με ποιον τρόπο δημιουργούν αξία ε, τα ε, τέτοιου είδου ψηφιακά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση ε, δεν υπάρχει συμφωνία σε ό,τι αφορά την ίδια τη διαδικασία δημιουργίας αξίας σε σχέση με τα ψηφιακά αγαθά. Ε, πράγμα το οποίο με φέρνει ε, στι 15 δράσεις κατά του BEPS από την πλευρά του ΩΣΑ. έχει υπάρξει αποτελεσματικό σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ελαχίστων προτύπων με αυτές τις 15 δράσεις. με, με κάποιες ουσιαστικές σε ό,τι αφορά ορισμένα φορολογικά καθεστώτα, σε ό,τι αφορά τι αναφορέ αναχώρα, και ο αντίκτυπος ορισμένων από τα μέτρα του ΩΣΑ είναι ορατός γιατί τα καθεστώτα διανοητικά ε, ιδιοκτησία σχετίζονται τώρα πλέον ε, στενά με τους κανόνες σε ό,τι αφορά την έρευνα και την ε, καινοτομία, ενώ υπάρχει και το ζήτημα των cashboxes. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτού του είδους οι τεχνολογίες που απαντώνται εδώ είναι ε, πολύ περίπλοκες και γι' αυτό είναι δύσκολο να αξιολογηθούν. Οι περισσότερε δράσει σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση δεν ε, σημειώνουν μεγάλη ε, πρόοδο. Για παράδειγμα δεν υπάρχει συμφωνία σε ό,τι αφορά την μόνιμη εγκατάσταση και τη δράση 7 δεν υπάρχει συμφωνία αλλά και η ε, αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων από τις δράσεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εθνικές νομοθεσίες. Ε, ωστόσο, οι καλές ειδήσει είναι ότι οι φορολογικές αρχές έχουν πλέον καλύτερα εργαλεία στη διάθεσή τους ε, για να διαπιστώνουν πότε λαμβάνει χώρα, η πρώτη, λαμβάνουν χώρα δραστηριότητε μετατόπισης των κερδών. Ε, επίσης, υπάρχουν και κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες εσκεμμένα και θελοντικά προβαίνουν σε μια ε, αναστήσα της δομές τους, ούτως ώστε να ε, ευθυγραμμίζονται με τις σχετικές ε, διατάξεις. Υπάρχουν και περαιτέρω νομοθεσίες ε, εδώ, για παράδειγμα, στις στην Ευρώπη, στην Κίνα και σε, άλλους, σε άλλες χώρες όπου εφαρμόζονται αντίστοιχοι κανόνες και σε ό,τι αφορά το απλουστευμένο σύστημα συμμόρφωση, το οποίο εφαρμόστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια των συστάσεων του ΩΣΑ οδήγησε πράγματι σε αύξηση των εισόδων κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα ωστόσο υπάρχουν πολλά μονομερή μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Γαλλία, ε, και το Ηνωμένο Βασίλειο και μετά έχουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, με, την, με το σχετική νομοθεσία σε ό,τι αφορά τη διάβρωση φορολογική βάση και την καταπολέμηση των καταχρήσεων, αλλά έχουμε και το Ισραήλ και την Ινδία με, τον σχετικό, με το σχετικό φόρο equalization. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν από τέτοια μέτρα, μπορούν να έχουν δηλαδή αρνητικό αντίκτυπο για τι επενδύσει, μπορούν να έχουν ε, αντίκτυπο ε, στην ε, καινοτομία και την ανάπτυξη, ενώ μπορούν να θέσουν να μετατοπίσουν ουσιαστικά το άχθος, το σχετικό άχθος στους καταναλωτές ενώ ε, μπορούν να προκύψουν και περαιτέρω να πάνε σε επίπεδο διοικητικό και σε επίπεδο συμμόρφωση. Ε, και ο ΣΑΝ αναφέρεται στην ανησυχία του σε σχέση με τον σχεδιασμό αυτών των μέτρων, τα οποία βέβαια προφανώ θα πρέπει να συμμορφώνονται με την διεθνή νομοθεσία, ε, αλλά και σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τι τέσσερι θεμελιώδει ελευθερίε, αλλά και μετά όσα προβλέπει η συμμετοχή σε διάφορου διεθνεί οργανισμού όπω ο ΣΑΝ. Επίσης ε, τα πρόχρονα αυτά τα συστήματα θα πρέπει να αναφέρονται στα βασικά στους βασικούς στα βασικά ζητήματα που θέτει ο σάι Για παράδειγμα, εδώ μπορούμε να αναφέρουμε τις ε, διαφημιστικές υπηρεσίες ε, στο διαδίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς ακολουθεί τη γενικότερη τάση, ειδικότερα με τις οδηγίες της 21ης Μαρτίου. Έχει ξεκινήσει δηλαδή μια συζήτηση σε ό,τι αφορά την ε, δίκαιη νομοθεσία. Γιατί βέβαια σε ορισμένε περιπτώσει έχουμε κάποιε επιχειρήσει οι οποίε ε, ε, καταβάλουν φόρου με φορολογικό συντελεστή μόνο τη τάξη του 1,5% ενώ ο κανονικό φορολογικό συντελεστή είναι 23%. Και αυτό βέβαια θέτει πιέσει στι αρμόδιε αρχέ των κρατών μελών. Και υπάρχουν βέβαια ειδικοί φόροι που εφαρμόζονται εδώ, ψηφιακού δηλαδή χαρακτήρα και οι οποίοι βασίζονται ε, στον κύκλο εργασιών, τον αριθμό των χρηστών ε, και επίσης προβλέπονται και κάποιες εξαιρέσεις. Όλα αυτά τα μέτρα ευθυγραμμίζονται με τις συστάσεις του ΩΣΑ και πράγματι εστιάζουν στις επιχειρήσεις οι οποίες ε, παρουσιάζουν τον υψηλότερο κίνδυνο για ΠΕΠΣ. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δεν ευθυγραμμίζεται με αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί λίγο από την πρόταση τη Επιτροπή το Κοινοβούλιο είχε προτείνει ε, ε, ένα σύστημα σε ό,τι αφορά την κοινή κατάσταση, το οποίο θα ε, μπορούσε να προσθεθεί στο εφιστάμενο CCCTB. Η Επιτροπή είπε ότι θα μπορούσε κάτι τέτοιο να επιβληθεί αργότερα στο CCTB επιπροσθέτω, αλλά βέβαια υπάρχει κάποια ανησυχία ω προ το τι θα συμβεί τελικά σε σχέση με αυτά τα ε, μέτρα στο μέλλον. Επίση, και το ίδιο το CCCTB αποτελεί ένα πρόβλημα για τα κράτη-μέλη, καθώ ορισμένα έχουν υψηλότερο και άλλα χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή. Οπότε σε μακροπρόθεσμα θα πρέπει να αποφύγουμε ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την επιβολή του χαμηλότερου φόρου. Και α μην ξεχνάμε βέβαια ότι υπάρχει διαφορετικό επίπεδο τεχνολογιών ανά τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν επίση ε, τεχνικά προβλήματα που δημιουργεί η πρόταση τη Επιτροπή. Καθώς υπάρχουν διαφορετικές, ε, υπάρχει διαφορετική φύση, αν θέλετε, των επιχειρήσεων στο τομέα των ψηφιακών αγαθών. Είναι δηλαδή πολύ διαφοροποιημένες. Υπάρχουν παραδοσιακέ επιχειρήσει οι οποίε ταυτόχρονα μπορούν να βρεθούν στο στόχαστο τέτοιου είδου αδιατάξεων. Ενώ ε, γίνεται πολλή λόγο για τι ε, μικρέ επιχειρήσει, γιατί αναφέρεται ότι για παράδειγμα δεν είναι θεμητό να επιβάλλει το ίδιο φορολογικό συντελεστή στους διαμεσολαβητές ε, ε, και τους ε, εκείνους για παράδειγμα που προβλήνουν στις online και σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να υπάρξει αντίκτυπος για τις μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δρούν ως online διαμεσολαβητές. Μάλιστα τέτοια μέτρα μπορούν να είναι αρνητικά μακροπρόθεσμα για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν επιθυμούν να μεγαλώσουν περαιτέρω και δεν επιθυμούν δηλαδή να ε, ξεπεράσουν το σχετικό κατόφλι που προβλέπει η Επιτροπή. Επίσης, ε, τα σχετικά δεδομένα ε, τα οποία μπορούν να συλλέγουν οι ευρωπαϊκές αρχές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των χρηστών. Επίσης, τίθεται το ζήτημα των πλαστών ταυτοτήτων και των bots και της εγκατάστασης συμπληρωματικού λογισμικού το οποίο παρακολουθεί τους χρήστες και το οποίο θέτει περαιτέρω ε, επιβαρύνσεις ε, για τους καταναλωτές. Εδώ βέβαια έχουμε διαφορετική, διαφορετικές απόψεις εντός της Ευρωπαϊκής Για παράδειγμα, οι ε, σκανδιναβικές χώρες λένε πως η επιβολή ενός τέλους φορολογικού σε ενιαίο βαθμό ουσιαστικά δεν ευνοεί εκείνους ε, που θέλουμε, ενώ αντιθέτα σε ε, κάποιες άλλες χώρες όπως η Σουηδία, η, η ε, Γαλλία, η Αυστρία και άλλες είναι υπέρ τέτοιου είδους διαφορών μεταξύ των κρατών Τώρα, αν δούμε την θέση της Γερμανίας, κατά τις τελευταίες εβδομάδες είδαμε ότι εξέφρασε έναν ε, φόβο σε ό,τι αφορά τα αντίπνα από την πλευρά των πολιτιών. Είδαμε για παράδειγμα τι έχει συμβεί σε επίπεδο αλουμινίου, εισαγωγών αλουμινίου και ε, προφανώς ε, οι αρμόδιοι για τη χάραξη της πολιτικής δεν θέλουν να υπάρξει ένας φορολογικός πόλεμος αν Οπότε δεν θέλουν δηλαδή να βρεθούν σε μια κατάσταση όπου θα υπάρξουν αντίπεινα η θέση των ΗΠΑ είναι πολύ σημαντική σε αυτό το πλαίσιο, γιατί οι ΗΠΑ δεν θέλουν να βάλουν στο στόχαστρο ειδικά τι ψηφιακέ επιχειρήσει. Επίση, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ε, πώ οι σχετικέ επιχειρήσει μεταβάλλουν ήδη τη δομή του ε, και μετά από την επιβολή τη νομοθεσία που εγκρίθηκε το 2017 ε, δεν θα χρειαστεί περαιτέρω μεταρρύθμιση του συστήματος. Είναι σημαντικό να ε, τονίσουμε εδώ ότι ο φορολογικό συντελεστή σημειώθηκε στο 21% στι ΗΠΑ το 2017 και υπάρχει ένα έντος επαναπατρισμού των σχετικών φορολογικών εσόδων αφού υπάρχει και το σχετικό κατόφλι του 10% μετοχών των ΗΠΑ σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στο εξωτερικό και ούτω καθεξής. Αυτές λοιπόν αλλαγές Αυτές οι αλλαγές σημαίνουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ουσιαστικά η αξία παράγεται στη δική τους επικράτεια και κατά συνέπεια η επιβολή της φορολογίας θα πρέπει να γίνεται εκεί. Προφανώς δεν υπάρχουν, υπάρχουν άλλα σε χώρες οι οποίες διαφωνούν με αυτήν τη στάση και υπάρχουν 113 χώρες οι οποίες εργάζονται επί των συστημάτων της ψηφιακής ε, φορολογίας. Ε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν πως νομοθεσία τύπου data nexus συν του BEPS, ε, χωρίς ε, δηλαδή να καλύπτεται πλήρως η ψηφιακή οικονομία. Ε, υπάρχει από εκεί και μετά μια άλλη ομάδα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Ένωση που επιθυμούν την λήψη πολύ πιο συγκεκριμένων μέτρων. Και επίσης θα πρέπει να δούμε τις νέες τεχνολογίες που στηρίζουν το blockchain, τεχνολογία των αντικειμένων και όλα αυτά τα τμήματα της ε, κατανεμημένης ε, οικονομίας που μπορεί και να ε, προξενήσουν ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες στη φορολογική αρχή στο μέλλον. Βέβαια πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, ως προς το, η στόχευση γιατί μπορεί και οι διεθνείς προσπάθειες μέσω όσα και λοιπόν διεθνών πλατφορμών να ε, γίνουν πιο δυσχερείς και μπορεί να αρχίσει και πόλεμος φορολογικός ούτως είναι ανταγωνισμός. Πρέπει να, λάβουμε πρέπει να προχωρήσουμε πολύ προσεκτικά. Δηλαδή, λαμβάνοντα υπόψη και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερη πρόοδο. Έχουμε το στόχο για συμφωνία το 2020 στον ΩΣΑ, αλλά θα ήταν καλύτερο βεβαίω σε παγκόσμιο επίπεδο να εξασφαλιστεί η συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ, Έλλη. Ο δεύτερο ομιλητή τώρα ο Τζον Βέλα από το Κέντρο για την Φορολογία Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδας. Ελπίζω να βλέπετε καλά τις ε, διαφάνειες εκεί. Αυτό που θα ήθελα να κάνω εγώ στην ε, παρουσίασή μου, αφού μας εξήγησε η Ελίζα πολύ καλά πώς έχει προχωρήσει η κατάσταση, είναι μια, να πάρω απόσταση και να σκεφτώ λίγο περισσότερο τα θέματα σε όρους πολιτικής που αντιμετωπίζουμε τώρα και προς τα πού μπορούμε να κινηθούμε ή όχι. Το Διεθνές Φορολογικό Σύστημα, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, το σύστημα φορολόγησης του διεθνούς επιχειρηματικού κεφαλαίου βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση. σε μια πολύ σημαντική συγκυρία και για τον εξή λόγο. Όπως είπε και η Έλλη, κάποιες χώρες έχουν διάθεση για μεταρρυθμίσεις, αλλά διαφωνούν σοβαρό προ τον τύπο των ε, μεταρρυθμίσεων που θα εισαγάγουν. Τρεις ομάδες χωρών μπορώ να ξεχωρίσω, οι, ομα, ομάδες ε, απόψεων. Η πρώτη ομάδα κρατών λοιπόν πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη για αλλαγή, αλλά μόνο στοχευμένη Πιστεύουν δηλαδή ότι η αλλαγή θα πρέπει να γίνει κατά τρόπον ώστε να στοχεύονται συγκεκριμένες ψηφιακές επιχειρήσεις, επιχειρήσει ψηφιακής οικονομίας. Μια άλλη σειρά, μια άλλη ομάδα χωρών πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη για αλλαγή, αλλά ε, πρέπει να αλλάξει όλο το φορολογικό σύστημα. Δηλαδή η αλλαγή αυτή πρέπει να ξεπεράσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ψηφιακέ επιχειρήσει αλλά να και να επεκταθεί σε ολόκληρο το φορολογικό σύστημα. Ε, τρίτη ομάδα χωρών αυτέ οι οποίε θεωρούν ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ουσιαστική μεταρρύθμιση και άρα η πιο σημαντική μεταρρύθμιση των του φορολογικού συστήματο την τελευταία εκατοτετηρίδα ε, που έγινε με τον ΠΕΠΣ του αρκεί και δεν χρειάζεται να προχωρήσουν περισσότερο. Κρίσιμη λοιπόν η φάση στην οποία βρισκόμαστε, δεν ξέρουμε ποιο θα επικρατήσει από τι τρει αυτέ ομάδε. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω θα μπορούσε να ενταχθεί στην πρώτη κατηγορία. στοχευμένε δηλαδή μεταρρυθμίσεις αφορούν ειδικά τις επιχειρήσεις με υψηλή ψηφιοποίηση και πολλά κράτη-μέλη υπάγονται σε αυτή την κατηγορία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι θα μπορούσε γενικά να ταξινομηθεί στη δεύτερη ομάδα. Δηλαδή το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι πρέπει οι αλλαγέ να αφορούν όλο το φορολογικό σύστημα και όχι μόνο την ψηφιακή οικονομία. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά τι θέσει του Κοινοβουλίου, σε αυτό ε, τάσομαι και εγώ. Πιστεύω δηλαδή ότι έχουμε σημαντική ευκαιρία, χάρη στην ψηφιοποίηση τώρα, να φέρουμε αλλαγέ καθολικέ στο σύστημα. Και ελπίζω πράγματι να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. Κάπου είχα προβλέψει εδώ μία παράθεση από την διάμεση έκθεση που δημοσιεύτηκε από τον ΩΣΑ το Μάρτιο του 2018 και αναφέρομαι στη δεύτερη ομάδα, άρα εκφράζονται και οι δικές μου θέσεις Λέει λοιπόν ότι η μεταμόρφωση της οικονομίας και γενικότερα των τάσεων που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση μπορεί να παρουσιάζει προκλήσεις ως προς την συνεχιζόμενη αποτελεσματικότητα της, του υφισταμένου διεθνού συστήματος ε, φορολογίας για το επιχειρηματικό κέρδος. Δηλαδή, αφενός μεν μας λέει ότι δεν μπορούμε να μιλούμε μόνο για ψηφιακή οικονομία γιατί ζούμε σε παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και άρα μιλούμε για ψηφιοποίηση όχι τη οικονομία ή τη επιχείρηση, αλλά ολόκληρης ε, ε, όχι μόνο μιας επιχείρησης ή δραστηριότητα, αλλά ολόκληρης της οικονομίας δεν έχει νόημα να κοιτούμε μόνο τα επιχειρήσεις υψηλής ψηφιοποίησης. Αφενός αφετέρου δε θα παρατηρήσετε εδώ ότι τα προβλήματα που εντοπίζονται για τη δεύτερη αυτή ομάδα δεν είναι προβλήματα που μόνο από την ψηφιακή μετάλλαξη της κοινωνίας αλλά περισσότερο με τις τάσεις που φέρνει η παγκοσμιοποίηση. Όπως είπα, προσωπικώς συμφωνώ και εντάσσουμε στη δεύτερη αυτή ομάδα. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια καθολική αλλαγή συστήματο και όχι μόνο για την ψηφιακή οικονομία. Αλλά εάν έχουμε μεταρρύθμιση, τι είδου μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει, αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται. Και νομίζω ότι καλό σημείο εκείνη θα ήταν να πούμε τι είδου μεταρρύθμιση θα πρέπει για να την ε, ε, περιγράψουμε τη μεταρρύθμιση αυτή, να επιλέξουμε την κατεύθυνση, να κοιτάξουμε ποια είναι η ρίζα του προβλήματος, τι κοιτούμε να αλλάξουμε να μεταρρυθμίσουμε, αν μπορούμε να εντοπίσουμε τη ρίζα του προβλήματος, τότε έχουμε και καλύτερη ευκαιρία για εισαγωγή μεταρρυθμίσεων που θα αντιμετωπίζουν το κακό στη ρίζα του. Η ψηφιοποίηση για μένα δεν γεννά νέα προβλήματα σε σχέση με το υφιστάμενο πρόβλημα. Απλώς διονγκώνει τα υφιστάμενα προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά τα επιδεινώνει σημαντικά. Πώς το καταφέρνει αυτό η ψηφιοποίηση. Το καθιστά δυνατόν μέσω μιας διαδικασίας διεθνοποίησης. Η ψηφιοποίηση συνδυασμένη με τη διεθνοποίηση επιτρέπει σε μια επιχείρηση να έχει δραστηριότητες ε, σε όλο τον κόσμο. Να απευθύνεται σε ε, κεφαλαιοκράτες, σε μετόχους, σε ολόκληρο τον κόσμο. Να αναπτύσσει τις δραστηριότητές της, την παραγωγή της, το marketing, τη διαφήμιση κτλ. σε όλο τον κόσμο και να απευθύνεται στον καταναλωτή σε ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ έχουμε την κυρία διαφορά που οφείλουμε στην ψηφιοποίηση και από την οποία πορεύουν μια σειρά επιπλέον προβλημάτων που θα εξηγήσω, τα οποία όμως πιστεύω ε, έχουν τη ρίζα τους σε ένα παράγοντα. Ότι στο υφιστάμενο σύστημα η επιχείρηση φορολογείται στην έδρα του ακίνητου τη έδρα τη, ενό ακινήτου, δηλαδή εκεί που θα δηλώσει την έδρα τη εταιρεία, εκεί που θα δηλώσει το, εκεί που θα έχει το IP, το Internet Protocol διεύθυνση και ούτω καθεξής. Έτσι ορίζεται ο τρόπος φορολόγησης των επιχειρήσεων και από αυτό απορρέουν μια σειρά από προβλήματα, εκ των οποίων σε τρία θέλω να σταθώ, αν μπορώ να κάνω να προχωρήσουν και οι διαφάνειες, μάλλον δεν δουλεύει το κουμπί. Τώρα δούλεψε. Πάλι δεν δουλεύει. Uh, no, back. Μήπως να βγάλετε εσείς τον κούρσορα από την οθόνη για να μπορώ εγώ να χρησιμοποιήσω το τέτοιο. <laughs> No, Okay. Can you just can you just upload the whole slide? No, forward. Yeah. <laughs> One back. Sorry. Yeah, this is going to be fun. Θα το γλεντήσουμε από ό,τι βλέπω. Μπρος πίσω, όχι. Στην επόμενη διαφάνεια... Ίσως έτσι θα ήταν και πιο εύκολο. Uh, yeah, perfect. Okay, so um, the point I was trying to make is that um, the existing system has, has had... Το εφιστάμενο σύστημα έχει εδώ και χρόνια προβλήματα. Με την ψηφιοποίηση γίνονται χειρότερα. Αν κοιτάξουμε λοιπόν τη ρίζα του προβλήματος σε έναν βαθμό, θεωρώ ότι υπό το υφιστάμενο σύστημα ε, η φορολόγηση των επιχειρήσεων ε, στοχεύει στο που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις. Με αυτό το σύστημα μπορούν οι επιχειρήσεις όμως να μετατοπίζουν το κέρδος με μια σειρά από γνωστές τεχνιο λογίες όπως σε παραδείγμα να ορίσουν το IP σε ε, φορολογικές έδρες χαμηλής φορολόγησης. Αυτό υπήρχε ήδη. Με την ψηφιοποίηση γίνεται χειρότερο. Και διανοηθείτε πόσο σημαντικό είναι το Internet Protocol ε, για μια ψηφιακή εταιρεία. Μετά, επειδή υπάρχει αυτό το φορολογικό σύστημα με εστίαση στην έδρα, μπορούν να μετατοπίζουν τις δραστηριότητες τους επιχειρήσεις στις ε, δικαιοδοσίες χαμηλή φορολογία, χαμηλού φορολογικού συντελεστή και σας ε, υπενθυμίζω ότι ε, ακόμα και μονάδες παραγωγικές μπορούν να είναι κινητικές για όρους, σε όρους φορολογικούς επειδή ακριβώς υπάρχει το σύστημα αυτό. Χάρη στην ψηφιοποίηση. Το τρίτο πρόβλημα είναι των δύο προηγουμένων. Επειδή ακριβώς έχουν αυτό το κίνητρο για μετατόπιση του κέρδους στις δικαιοδοσίες χαμηλό φορολογικής βάσης και αντίστοιχα των ε, δραστηριοτήτων τους, έρχονται οι χώρες τώρα να υποχρεωθούν να μειώσουν την φορολογική βάση για να προσελκύσουν αυτές τις εταιρείε. Και αυτό ε, αποδυναμώνει το σύστημα, το αποσταθεροποιεί και θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά του μακροπρόθεσμα. Τώρα τι γίνεται λόγω αυτών των ε, ανταγωνιστικών πιέσεων, βλέπουμε μια μειωτική τάση στην φορολογική βάση των επιχειρήσεων, η οποία μειούται σταθερά τα τελευταία χρόνια, είναι σαφής η τάση στις G20, στις χώρες του G20. βλέπετε σταθμισμένο και μη σταθμισμένο μέσο όρο της ε, επιχειρηματικής φορολογικής βάσης αναλογά στις χώρες αυτές, μέσο όρο. Και νομίζω ότι απλώς μια τάση την οποία είχαμε πριν από την ψηφιοποίηση δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να επιβεβαιώνεται χάρη στην ψηφιοποίηση και να εντείνεται. Η κατεύθυνση είναι μία από ό,τι βλέπουμε και έχουμε λόγους να ανησυχούμε. Εάν λοιπόν δεν μπορούμε να βρούμε κάποιο τρόπο να το σταματήσουμε ή μάλλον εάν δεν έχουμε κάποιο λόγο να το σταματήσουμε αρκετά σοβαρό και δεν βλέπω να υφίσατε τέτοιου λόγο λόγος σοβαρός μέσα στο σύστημα, ένα σύστημα δηλαδή αυτόματο, δεν θα μπορέσει να σταματήσει αυτή η τάση. Η ψηφιοποίηση λοιπόν. Δεν γεννά νέα προβλήματα για μένα, απλώς τα επιδεινώνει λύση. Τι λύση μπορούμε να προτείνουμε. Εάν το πρόβλημα είναι μια από τις βασικές ε, πηγές του προβλήματος είναι το ότι επιδιώκει να ορίσει έδρα ε, εκεί που έχει τις κινητές αξίες μια εταιρεία, το φορολογικό σύστημα, θα πρέπει να αλλάξει αυτό το κριτήριο, δηλαδή να φορολογείται η έδρα η εταιρεία εκεί που η έδρα της έχει τα ακίνητα περιουσιακά της στοιχεία, τα οποία εξ ορισμού δεν αλλάζουν. Επιλογές. Πού βρίσκονται οι καταναλωτές της ή πού βρίσκονται οι μέτοχοι της εταιρείας. Προορισμός ή προέλευση δηλαδή, η καταγωγή της επιχειρήσης. Ας κοιτάξω τον, τον προορισμό ως λύση, μια και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εάν ορίσουμε ως βάση τον προορισμό, για το προσδοσμό τη φορολογική ε, έδρα. Λύνονται και τα τρία προβλήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε κανένα άλλο πρόβλημα. Δεν είναι ότι έχουμε βρει την πανάκια, ότι δεν θα έχουμε καμία δυσκολία. Φυσικά και θα υπάρξουν δυσκολίε. Αλλά βλέπω να υπόσχεται πολλά αυτή η λύση μακροπρόθεσμα, ιδιαίτερα εάν, όπω εγώ, πιστεύει κανεί ότι είναι μη βιώσιμο μακροπρόθεσμα το υφιστάμενο σύστημα. Τώρα, μπορεί πριν από μερικά χρόνια να φαινόταν ε, πολύ αμφιλεγόμενο και να προξενούσε μεγάλες αντιδράσεις ε, το επιχείρημα του στοιχείου της, ε, του προορισμού ως επιλογή της φορολογικής βάσης. Τώρα πια αυτό έχει ξεπεραστεί και άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα εκεί κινείται. Αλλά αυτό που θα ήταν λάθος θα ήταν με τις αρχές που έχουμε αυτή τη στιγμή να επιβάλλουμε μόνο το σύστημα του προορισμού. Ε, δηλαδή πηγή έδρα και επιπλέον αυτού να επιβληθεί και η έννοια του προορισμού της δραστηριότητας της επιχείρησης. Αυτό θα ήταν λάθος. Γιατί θα οδηγούσε σε περισσότερη ασάφεια στο σύστημα και άρα εγώ πιστεύω ότι θα ήταν πολύ προτιμότερο αντί να γινόταν αυτό να προχωρούσαμε προς ένα σύστημα το οποίο συνολικά με συνέπεια έδινε ως βάση φορολογική το σημείο προορισμού της επιχειρηματική δραστηριότητας μιας εταιρείας. Με διάφορους τρόπους μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό μπορούμε να περάσουμε σε ένα καθαρό αμυγέ σύστημα προορισμού. Υπάρχει δυνατότητα σε ακραία συστήματα όπως ο φόρος ε, ρευστότητας η κίνηση του χρήματος που είναι για μένα ο καλύτερος αλλά και άλλα τα οποία ίσως πολιτικά να μην είναι όμως τόσο εύπεπτα και άρα μπορούμε να κοιτάξουμε μια συνολική και συνεπή λύση για την επιλογή του προορισμού ως βάση για τη φορολογία, χωρίς όμως να φτάσουμε στα αμυγή συστήματα. Τα, από συστήματα λοιπόν αυτά που έχουν προτείνει η Αβιγιόναχ, Κλάουζινγκ, Durst, Schreiber και Fell και άλλοι υπό τον Μάικ Τέβερον, τον οποίο και δεν υποστηρίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια τέτοια πρόταση, άλλοι καθηγητές είναι αυτοί. Τι κάνουν λοιπόν, προσπαθούν κάποιο από το φορολογητέο έσοδο να το εντοπίσουν σε μια χώρα της δραστηριότητας και το υπόλοιπο ποσό να το αναγάγουν σε μια χώρα προορισμού. Δηλαδή ένα κομμάτι από την πίτα θα το πάρει η χώρα της δραστηριότητας, αλλά πάλι τα ωφέλη σε σχέση με τον προορισμό ε, του προϊόντος ε, θα φορολογηθούν στη χώρα του προορισμού. Στο μεγαλύτερό τους ποσοστό. Δηλαδή, εάν τώρα τίνουν οι χώρες, οι επιχειρήσεις, να εξασφαλίσουν, μάλλον οι χώρες τίνουν να φορολογούν ε, τα τακτικά έσοδα που προκύπτουν από τακτικές ε, δραστηριότητες, δηλαδή το προϊόν που παράγει και πολύ μια ε, επιχείρηση με εργοστάσιο, δεν βλέπει, δεν καλύπτει το σύστημα τώρα αυτό το οποίο θα μπορούσε να είναι μια διαφορετική προσέγγιση, δηλαδή όχι το τακτό έσοδο. Γι' αυτό λέμε ας αφήσουμε εκεί που είναι τα τακτά έσοδα, αλλά το υπόλοιπο αντί να μπορεί να το μεταφέρει σε ένα φορολογικό παράδεισο ή σε μια χώρα χαμηλής φορολόγησης, ας το φορολογήσει η χώρα προορισμού. Με αποτέλεσμα βέβαια κάποια στιγμή και από την προοπτική των χωρών μελών αναλόγως να έχουμε κερδισμένους και χαμένους αν αυτό το σύστημα αυτό, αλλά τουλάχιστον έχουμε λύσει το πρόβλημα που σας ανέφερα και νωρίτερα, Το αν είναι βιώσιμο το σύστημα μακροπρόθεσμα, γιατί πράγματι δεν έχουμε επιλογή σε αυτό. Εδώ έχουμε ένα σύστημα που είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα και νομίζω ότι ενώ τα προβλήματα προϋπήρχαν, η ψηφιοποίηση μας αναγκάζει να τα δούμε πολύ πιο σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ καθηγητά Βέλα για τα όσα μας ε, είπατε. Και τώρα γύρω στον ερωτήσεων από πλευρά των βουλευτών σύμφωνα με τη λίστα ο υποφαινόμενος που είναι ο συνεισηγητής. Έχω ερωτήσεις και για τους δύο. Ξεκινώ από τον δεύτερο, τον κύριο Βέλλα. Να καταλάβω καλύτερα το αναθεωρημένο φορολογικό σύστημα το οποίο πρεσβεύεται. Για πέστε μας λίγο περισσότερα με ένα πρακτικό παράδειγμα. Η Facebook, η Apple, τι θα γινόντουσαν αν υπήρχε ένα τέτοιο σύστημα. Τι σύστημα θα τις δείπε επίσης. Τι γίνεται με το συντελεστή εταιρικού φόρου και το σύστημα επί τη της χώρας. Είχαμε έναν κοινό φοροσοδήματος, αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τα κρατημέλη. Κοινό μέτωπο. Να συνδεθεί επομένω αυτό το κοινό μέτωπο φοροσοδήματος με τον εταιρικό φόρο. Ναι, ναι, θα ε, σας πω για τη δεύτερη ερώτηση, είναι πιο εύκολη. Πρώτα, πρώτα. Είναι το θέμα πολιτικό. Αν ποτέ θα συμφωνήσουν τα κρατη να υπάρχει μια τέτοια φορολογική βάση για εταιρικό φόρο. Και σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται. Όταν ε, κάποια χρόνο που δεν συμφώνησε έχει πιο χαμηλό φόρο, οπότε έχουμε μετατόπιση, φυγή των εταιριών εκεί που έχουμε μικρότερη φόρη. Πρόεδρος. Ναι, αλλά ήθελα να πω κάτι άλλο. Αν υπάρχει ε, αυτή η κοινή βάση, δεν θα ήταν περιθώριο για να υπάρξει ένα κοινό σύστημα. Τελικά. Έτσι θα είχαν το, περιθώριο, το χρονικό περιθώριο τα κρατημέλη να προχωρήσουν προς ένα κοινό νέο σύστημα βέλα. Όχι, ποτέ δεν υποτίθεται σε μια πενταετία θα, θα καταρρεύσει το σύστημα του εταιρικού φορού, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό. Νομίζω έχει ενίο συντελεστή ψηφιακό του μάλλον ε, ενίο συντελεστή ενός ψηφίου, μονοψήφιο, η Ουγγαρία. Άρα, Ναι, θα, θα υπήρχε το περιθώριο να προβληματιστεί κανείς για κάποια μεταρρύθμιση πριν έχουμε κατάρρευση του συστήματος. Αν υπάρξει συμφωνία. Ναι, αυτό θα ε, έδινε χρόνο. Υπάρχει, υπάρχει ο χρόνος. Για την πρώτη σας ερώτηση τώρα. Ένα παράδειγμα εκτός των ψηφιακών. Αν θεωρήσουμε μια εταιρεία. Έχει στη χώρα Α ένα εργοστάσιο, κάνει το marketing στη χώρα Β και πουλάει και στην χώρα Α και στη χώρα Β και σε μια χώρα Γ. Και επειδή υπάρχει εταιρική δραστηριότητα στην Α και στη Β χώρα, το σύστημα λέει ναι, ας φορολογηθεί εκεί. Γιατί εκεί έχει κέρδη. Όμως, τι γίνεται με το υπόλοιπο κέρδος που δεν θέλουμε καταλήξει σε φορολογικό παράδοσο. Τι είναι λοιπόν με αυτό το παραπάνω για κέρδος πέραν του συνήθους. Γι' αυτό λέμε κατανομή φορολογητέων κερδών ανάλογα με τις πωλήσει. Τι που τελικά πρέπει να θεωρηθεί ότι βρίσκονται οι καταναλωτέ των προϊόντων μια εταιρεία. Και έτσι να γίνει η κατανομή. Ο πολιτική πλευράς τώρα, ίσως αυτό, είναι πιο εύκολο να περάσει παρά η χώρα προορισμού αποκλειστικά σαν κριτήριο. Ευχαριστούμε καθηγητά λέει ο πρόεδρος. Ε, τώρα για σας ε, είπατε για Ιταλία, Γαλλία, ΙΠΑ, διάφορες χώρες. Όλες έχουν κάποιο ειδικό φόρο, ειδική φορολόγηση για τα ψηφιακά, κύριε Χατζήβα. Και στα πλαίσια της κουβέντας μας θα μπορούσαμε στην Ένωση κάτι να κάνουμε χωρίς να θεσπιστεί κάποιο κοινό πρότυπο. Χωρίς να υπάρχει τόση πανσπερμία μέτρων. Ε, ναι, τα ε, μέτρα του κάθε κράτους είναι πιο κακά για το εμπόριο όπως ας πούμε είπαμε για τον blockchain θα μπορούσε η Ένωση κάποια στιγμή να προτυποποιήσει αυτά τα μονομερή μέτρα γιατί πολλές φορές όπως και για την Ουγγαρία μπορεί να θεωρηθούν αυτά κρατική επιδότηση, ενίσχυση και σύμφωνα με τον ΟΣΑ όλα αυτά βασίζονται σε κάποιες αρχές δηλαδή όπως το BEPS της εταιρεία ε, ψηλότερου κινδύνου. Όπως η διαφήμιση, οι υπηρεσίε δημοσιολάβηση, εκεί υπάρχει υψηλότερο ρίσκο. Οπότε η πρωτοποίηση θα βοηθούσε από την άλλη μεριά. Μονομερή μετά τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελούσαν πάλι αντίπεινα και θα έφυγαν το σύνολο του συστήματος και μακροπρόθεσμα θα έπρεπε να βρεθεί κάποια λύση στα πλαίσια του ΟΣΑ σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ, λίγο Πρόεδρο, και πάμε τώρα. Θα που έχουν ζητήσει το λόγο τα πολιτικά κόμματα και το κυρία Ντανούτα Γεσλοβιέτσκα. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να υποβάλω την ερώτηση από πλευρά του συντονιστή του ΕΛΚ που δυστυχώ δεν μπόρεσε να παραστεί. Σα ευχαριστούμε πρώτα-πρώτα που ήρθατε και μα τα είπατε Και θέλω να ρωτήσω κάτι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τους δύο καλεσμένους μας. Όλοι εμπιστώνουμε ότι χρειάζεται δικαιώτης δικαιοσύνη στην επιβολή της φορολογίας ιδίω όσον αφορά τις ε, εταιρείε που ασχολούνται με τα ψηφιακά. Αυτό είναι λογικό στο πλαίσιο ψηφιακής οικονομίας. Τι γίνεται σε διεθνές επίπεδο. Τι γίνεται στα πλαίσια του ΩΣΑ και του G20. Αρχικά η Επιτροπή ήθελε να εστιαστεί σε αυτά τα διεθνή όργανα όσον αφορά την ψηφιακή φορολογία αλλά χωρίς να παραβλαβούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες. και θα μπορούσαν επίση να φυγούν οι εταιρείε ε, μακροπρόθεσμα. Τώρα έχουμε μια πολωνική εταιρεία, ονομάζεται Allegro και ανταγωνίζεται κάποιου πολυεθνικού, κάποιου διεθνεί ε, γίγαντε. Και τώρα αυτή η πλατφόρμα πρόκειται να φορολογηθεί Θα υποστεί πέραν του συνήθους φόρου και τον ψηφιακό φόρο. Αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποια εταιρεία σε οποιοδήποτε κράτο μέλο. Και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώ θα μπορούσε κανεί να αποφύγει το να Έχει καταλογιστεί κάποιο φόρο και να μπορέσει κάποια ευρωπαϊκή εταιρεία να συνεχίσει να δρά και να επενδύει. Ευχαριστούμε για την ερώτηση, αλλά δεν ήρθε ακόμα προ του Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, σε λίγο, σε λίγο. Αλλά δεν έχει σημασία, θα το λάβουν υπόψη να απαντήσουν προσκεκλημένου, την κύριε Χατζήβα. Ναι, αναφέρθηκα σε αυτά τα προβλήματα στην ε, εισήγηση Μα Βέβαια και θα θυγούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες από τέτοιο φόρο. Ιδίως οι μικρότερες επιχειρήσεις θα δυσκολευτούν να βρουν συγκριτικό πλεονέκτημα εάν το κόστος της διαφήμισης, ε, οι ε, προς τους καταναλωτές ε, αυξηθούν όσον αφορά το και η ισορροπημένη προσέγγιση είναι το καλύτερο. Δηλαδή, να μην κόψουμε τους πρωταθλητές μας Έχουμε Ευρωπαϊκή Εταιρεία στο τόπικο, των εταιρεών και αν θέλουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις θα πρέπει να βοηθήσουμε την κοινοτομία τους, την πρόοδο και άρα η φορολογία θα δημιουργήσει πρόβλημα. Πώ θα συνεχίσουν ανταγωνιστικέ με με επίπεδο ευρωπαϊκέ εταιρείε. Τώρα, μήπω θέλει να συμπληρώσει ο συνάδελφο Βέλα. Δεν θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να επιβληθεί φόρος για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Για πολλούς λόγους. Επιβάλλεται στον τζίρο μιας επιχείρησης, ούτω ώστε να εξισορροπηθεί η κατάσταση αν δεν υπάρχει φόρος επί των κερδών. Υπήρξε πρόταση για προσωρινή επιβολή. Μα ούτε αυτό όμως ε, είναι το καλύτερο και, η ίδια η Κομισιόν σε κάποια γραφό το έχει παραδεχτεί ότι δεν είναι η πιο καλή λύση. Ο πρόεδρος. Ευχαριστώ και προχωράμε. Σοσιαλδημοκράτε. Εύελιν Ρέγκνερ. Ευχαριστώ. Έχω κάνα δύο ερωτήσεις, καταρχάς προς τον καθηγητή Βέλα. Πολλά από αυτά τα οποία Έχουμε εμείς ορίσει και ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα διάφορα public CBCR, το ψηφιακό κέντρο δραστηριοτήτων κτλ. Ένα ερώτημα λοιπόν, πολιτικής φύσεως μάλλον. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσο μέσο πίεσης, μοχλός πίεσης προς τις Ηνωμένε Πολιτείες το θέμα της φορολογίας των ε, ψηφιακών επιχειρήσεων. Και δεύτερη ερώτηση. Είναι δυνατόν να την πρόταση της Επιτροπής κάποια επιχείρηση να έχει όλη την οικονομική της δραστηριότητα online καταχωρημένη. Δηλαδή, η συγχώνευση, η διέρεση, η κατανομή κτλ. Μπορεί να περνάνε όλα από ένα ψηφιακό αρχείο. Μπορεί να υπάρξει μια πλήρης ψηφιοποίηση της οικονομίας, γιατί ξέρουμε ότι σε ορισμένες χώρες λειτουργεί σωστά αυτό το σύστημα. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε δύο στοιχεία. Αφενός μεν την κινητικότητα των επιχειρήσεων, αφετέρου δε την ψηφιακή ίδρυση ή μεταμόρφωση. Και εδώ είναι η ερώτησή μου, γιατί έχει και νομικές συνέπειες. Σε ποιο βαθμό θα είναι καλύτερο ή χειρότερο ή πού πρέπει τέλος πάντων να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής και βέβαια το κίνδυνο να ιδρυθούν εταιρείες ε, γραμματοθυρίδες οι βιτρίνες. Όλα αυτά πώς μπορούν δηλαδή στην πράξη να υλοποιηθούν. Καταρχήν ο καθήτης Ναι, ήταν αρκετά εντελεχή η ερωτήση σα, οπότε θα προσπαθήσω να δώσω μια πλήρη απάντηση. Αν δεν τα καταφέρω, μπορείτε να, το θυμάστε. Καταρχήν, το πρώτο ερώτημα ήταν πολιτική φύση. Δηλαδή, πώς αυτό θα έχει ένα αντίκτυπο σε αυτό που φοβούνται πως εξελίσσεται, που φοβάται ο κόσμος πως εξελίσσεται σε έναν εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Πολιτείες. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις η αίσθηση που έχει ο κόσμος είναι ε, εξίσου σημαντική με την πραγματικότητα. Και η αίσθηση που υπάρχει σήμερα είναι ότι υπάρχει ένας εμπορικός πόλεμος. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, δηλαδή υπάρχει μια δυσαρέσκεια από την πλευρά των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την ε, υποστήριξη από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το βασικό πρόβλημα, κατά δική μου άποψη, είναι το εξή. Ανάμεσα στο 2013 έως 2015 ε, είχε ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση σε σχέση με το BEPS ε, και ε, το ζητούμενο εδώ δεν ήταν να γίνει μια ανακατανομή των δικαιωμάτων φορολόγηση μεταξύ των ε, κρατών ε, Και αυτό που έλεγε ο ΩΣΑ το, το διευκρίνησε ακριβώ αυτό. Δηλαδή το ΜΠΕΠΣ δεν έχει να κάνει με την ανακατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων. Υπάρχει απλώ μια πίτα εντό εισαγωγικών και θα πρέπει να δούμε πώ θα γίνει η κατανομή τη. Ακριβώς τώρα λοιπόν το πράγμα αρχίζει να γίνεται πιο επίκαιρο και πιο δύσκολο και από πολιτική άποψη, γιατί ακριβώ τίθεται το ερώτημα που σε αυτή την κατανομή τη πίτα ποιο θα πάρει πόσο μεγάλο κομμάτι. Ε, τώρα, αν κατάλαβα σωστά το ερώτημά σα και μπορείτε να με διορθώσετε στη συνέχεια, είναι το κατά πόσο είναι πρόβλημα το να προσπαθήσουμε να θέσουμε συγκεκριμένα όρια στην ψηφιακή οικονομία. Δηλαδή, μήπω οι μακροπρόθεσμε λύσει που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργούν ένα είδος περιχαράκωσης, ένα είδος οριοθέτησης γύρω από την ψηφιακή οικονομία. Κατά τη δική μου άποψη, ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Γιατί εδώ οι ορισμοί ε, ακριβώς ε, εστιάζουν και οι σχετικές λύσεις στο τι ακριβώς είναι μια ψηφιακή υπηρεσία, τι είναι ένα ψηφιακό αγαθό και θα χρειαστούν αυτά ούτε ώστε να γίνει η, η, ο επιμερισμός ε, του ενός ε, κέρδους σε μια συγκεκριμένη μόνιμη κατάσταση. Όμως όπως ήδη αναφέρθηκε τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε αν θέλουμε να έχουμε δόσμους θα πρέπει να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες οδηγίες ως προς το πώς θα γίνεται ο επιμερισμός συγκεκριμένου κέρδου σε μια συγκεκριμένη μόνιμη κατάσταση. Για παράδειγμα, αν υπάρξει σε δύο-τρία χρόνια μια νέα ε, ψηφιακή καινοτομία, τι θα σημαίνει αυτό. Θα πρέπει να αναθεωρηθούν ή να αναθεωρούνται δύο-τρία χρόνια όλοι οι σχετικοί κανόνες και όλη η σχετική καθοδήγηση. Δεν είμαι βέβαιος κατά πόσο ε, έχει νόημα να ακολουθήσουμε μια τέτοια πολιτική, συνεχών δηλαδή αναθεώρηση. Ευχαριστώ. Και ε, τώρα ε, η τελευταία στιγμή τη συζήτητρια, η κυρία Νίνα Αγγίλα για του Σοσιαλιστέ. Σα ευχαριστώ για την παρουσίασή σα Εστιάσαμε ιδιαίτερα στι Ηνωμένε Πολιτείε. Και προφανώ υπάρχουν πολλέ ψηφιακέ επιχειρήσει οι οποίε ε, έχουν την έδρα του εκεί, αλλά υπάρχουν άλλε τώρα που έχουν την έδρα του στην Κίνα. Οπότε το ερώτημα είναι πώ θα αντιδράσει η Κίνα στο σκεπτικό που ακολουθούμε εδώ με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και από εκεί και μετά, βέβαια, ο φόρος στον οποίο αναφερόμαστε είναι τελικά έμεσος και όχι άμεσος. Γιατί βέβαια αν είναι έτσι οι Ηνωμένε Πολιτείε οι οποίε υποστηρίζουν τον άμεσο φόρο ε, θα δημιουργήσουν πρόβλημα και θα υπάρξει πρόβλημα στο επίπεδο της σύσπραξης αυτών των φόρων. Ε, και βέβαια πριν από κάποιες εβδομάδες βρέθηκε εδώ ο Μάρκ Ζούπεργκερ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όταν του τέθηκε μια ερώτηση σε ό,τι αφορά την καταβολή φόρων μας είπε ότι καταβάλουμε τους φόρους μας όπου είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Οπότε ε, σας ρωτώ κύριε καθηγητά, εάν μπορέσουμε να φεύγουμε τα προβλήματα σχέση με την έσπραξη των φόρων, πού εντοπίζονται τα μεγάλα προβλήματα ως προς το να αναγκάσουμε τις ε, μεγάλες αυτές επιχειρήσεις να μην φοροδιαφεύγουν πλέον. Ευχαριστώ κύριος Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημά σας, ε, δεν γνωρίζω ποια θα είναι η αντίδραση της Κίνας. Δεν έχω διαβάσει κάτι σχετικά. Αλλά το ενδιαφέρον κομμάτι εδώ είναι το εξή. Οι Ηνωμένε Πολιτείε συμπεριλαμβάνονται στη δεύτερη ομάδα. Δηλαδή, μία ομάδα η οποία είναι διατεθειμένη να γίνουν ε, αλλαγές στο σύνολο του συστήματος, όχι μόνο στις ε, κατεξοχήν ψηφιοποιημένε επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν κατά κάποιο τρόπο οι Ηνωμένε Πολιτείε, κατά τη δική μου τουλάχιστον άποψη, υιοθετούν τη σωστή στάση ω προ το είδο τη μεταρρύθμιση που χρειαζόμαστε. Δηλαδή, συμφωνώ με την, ε, με την ε, ε, στάση εδώ που υιοθετεί η Αμερικανική πλευρά και την προτιμώ σε σύγκριση με αυτή που υιοθετούν ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή με την πρότασή τη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο στήριο τη ερώτησή σα, ως προς τις μακροπρόθεσμες λύσεις, ναι, υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την, την, την έννοια της μακροπρόθεσμης λύσης. Η μακροπρόθεσμη λύση ε, ε, ε, εδράζεται στο ότι θα πρέπει να φορολογούμε εκεί όπου δημιουργείται η αξία. Και στο σχετικό έγγραφο το οποίο εκπώνησε το τελευταίο Νοέμβριο η Επιτροπή αναφέρει η ίδια ότι είναι πολύ δύσκολο να διαπιστώσει κανείς το πού και πόση αξία παράγεται στον ψηφιοποιημένο κόσμο. Οπότε το ερώτημα που θέτω εγώ είναι το εξής. Εάν θεωρούμε πως είναι πολύ δύσκολο έστω και ποση αξια παραγεται στον ψηφιοποιημενο κοσμο οποτε το ερωτημα που θετω εγω ειναι το εξης εαν θεωρουμε πως ειναι πολυ δυσκολο εστω και να δούμε πού και πόση αξία παράγεται, τότε γιατί θεωρούμε σκόπιμο το να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο ακριβώς βασίζεται σε μια έννοια την οποία δεν μπορούμε να, να ορίσουμε ε, επακριβώς. Οπότε, πρωτού περάσουμε στο ζήτημα της συζήτησης σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του συγκεκριμένου φόρου, πρέπει να ε, δούμε το πόσο ανησυχητικό είναι και για μένα κατευθείαν δηλαδή χτυπάει εδώ ένα καμπανάκι το να μην γνωρίζουμε το, την βασική αρχή στην οποία θα βασίζεται αυτό το σύστημα. Άρα λοιπόν θα έχουμε εδώ εκτενείς κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα προσπαθούν να εξηγήσουν το πού ακριβώς παράγεται η αξία στις διάφορες αλυσίδες παραγωγικές αξίας αλλά ε, η ανησυχία μου είναι ότι καθώς τα πράγματα κινούνται τόσο γρήγορα αυτές οι οδηγίες πάντοτε αυτά είναι παροχημένες. Θα βρίσκονται πίσω από τα πράγματα. Άρα λοιπόν υπάρχουν και τεχνικά προβλήματα αλλά και σε ενιολογικό επίπεδο η πρόταση έχει βασιστεί σε, μια αρχή η οποία είναι αυτή καθ' αυτή προβληματική. Ναι, να προσθέσω και εγώ κάτι ε, στο ερώτημα που τέθηκε στον καθηγητή Βέλα ό,τι αφορά την Κίνα. Ε, θεωρώ πως η Κίνα ε, βρίσκεται σε ένα ψηφιακό, σε μια ψηφιακή φούσκα, δηλαδή είναι ψηφιακά απομονωμένη, γιατί ακριβώς έχει το δικό της Google, το δικό της Facebook, όπως δηλαδή και η Ρωσία. Αντιθέτω, οι αμερικανικέ επιχειρήσει ε, είναι δικαιωμένε και αξιοποιούν τα δικά μα δεδομένα, των δικών μας ε, χρηστών και γι' αυτό υπάρχει αυτή η άμεση και σημαντική συσχέτιση η δική μας με τις ΗΠΑ και γι' αυτό θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα μέτρα που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ. Και σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημα που θέσατε, σε ό,τι αφορά την καταστατήρηση του συστήματο, αυτέ οι έμενε, αυτέ οι επιχειρήσει πάντοτε βρίσκουν κάποια παραθυράκια στην νομοθεσία. Ε, πάντοτε προβλέπονται κάποιε εξαιρέσει και πάντοτε θα βρίσκουν κάποιου φορολογικού συμβούλου οι οποίοι θα βρίσκουν κάποια, κάποιο τρόπο να αποφύγουν την φορολόγηση και θα είναι και πολύ εφευρετικοί στο να το κάνουν αυτό. Όπως είπε ο Τζον, εξελίσσονται αυτέ οι ψηφιακέ τεχνολογίε τόσο γρήγορα έτσι ώστε οι φορολογικές αρχές να δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν αυτήν την ταχύτατη εξέλιξή τους. Οπότε αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Η Δανούτα από το ΕΛΚΑ θα θέσει το τελευταίο ερώτημά στους ομιλητές. nowego systemu opodatkowania. Κύριε Πρόεδρε, μας είπατε για κάποια λύση θεωρητικά. Είναι λογικό αυτό που είπατε. Άρα θα έπρεπε να πληρώνετε εκεί που έχει την έδρα της εταιρεία, στον τόπο κατοικίας όπως λέμε με το ένα σενάριο. Το άλλο σενάριο είναι για τον, στον τόπο προορισμού. Οπότε ως καταναλωτής απορώ μήπως δεν θα υπάρχει έτσι ανταγωνισμός και άρα τα αγαθά, αν κάποιο με πιο ψηφοφόρο θα φτάσουν αργότερα ή δεν θα φτάσουν καθόλου. Και δεν λέω για ψηφιακέ υπηρεσίε, λέω γενικώ για εμπορεύματα. Δεν υπάρχει αυτό ο κίνδυνο. Ε, καθηγητά Βέλα, νομίζω πως σε εσά απευθύνθηκε το ερώτημα. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να εξηγήσω ακριβώ αυτή την πρόταση. Πάντω, με βάση αυτή, ο φόρο δεν θα εφαρμόζεται με βάση τον τόπο κατοικία, αλλά με βάση το που λαμβάνει η χώρα η φορολογούμενη δραστηριότητα. Νομίζω πως το βασικό σας ερώτημα είναι τελικά το ποιο ε, τελικά είναι εκείνο ο οποίο επιβαρύνεται με τον φόρο. Δηλαδή, οι μέτοχοι θα είναι εκείνοι, οι εργαζόμενοι θα είναι εκείνοι που θα επιβαρυνθούν με τον φόρο ή για παράδειγμα οι καταναλωτέ μέσω αύξηση των ε, σχετικών τιμών. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ε, τελικά το ποιο είναι εκείνο ο οποίο επιβαρύνεται με τον ε, φόρο επιχειρήσεων. Ε, σίγουρα δεν είναι ίδιες επιχειρήσεις, οπότε γνωρίζουμε ότι όταν επιβάλλουμε ένα φόρο σε μια επιχειρήση γνωρίζουμε ότι δεν θα είναι εκείνη η οποία θα επιβαρυνθεί αλλά θα είναι κάποιο φυσικό πρόσωπο και γι' αυτό λέμε ότι θα είναι είτε οι μέτοχοι είτε οι εργαζόμενοι είτε οι καταναλωτές. Οπότε θεωρούμε πω προβληματική αυτή την έννοια του να γίνεται λόγο για φορολογία επιχειρήσεων, γιατί οι επιχειρήσει δεν καταβάλουν οι ίδιες αυτόν τον φόρο, είτε δηλαδή ε, θα μεταφερθεί στους μετόχους μας των μετοχών, είτε θα υπάρξει μείωση των μισθών, είτε θα υπάρξει αύξηση των τιμών των προϊόντων για του καταναλωτές. Οπότε δεν μπορώ να σας δώσω μια απάντηση σε σχέση με το τελικά ποιο θα επιβαρυνόταν με αυτόν τον φόρο στην πραγματικότητα με βάση αυτή την πρόταση. Και δεν έχουμε επαρκή στοιχεία στη διάθεσή μας ως προς το ποιος τελικά επιβαρύνεται και το με τον φόρο ε, επιχειρήσεων ο οποίος επιβάλλεται σήμερα στο σημερινό σύστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να κλείσουμε λοιπόν. Και να πω και εγώ δύο λόγια. Το τελευταίο σημείο που αναφέρατε για το τελικό κόστος του φόρου επιχειρήσεων είναι ένα ολόκληρο θέμα συζήτηση. Αλλά βεβαίω όταν υπάρχει διαφορετική φορολόγηση για τις εταιρείε ενό κλάδου ή γενικά τι επιχειρήσει, ε, έχουμε πρόβλημα ανταγωνισμού και βέβαια υπάρχει και θέμα εθνική δικαιοδοσίας, η οποία όμως χάνεται στη σύγχρονη εποχή. Η δικαιοδοσία για την επιβολή του φόρου, λόγω της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε το εξής, εάν ο μέτοχος γίνει το επίκεντρο της φορολογίας. Αυτή η κατανομή κέρδος που θα κατανέμεται μεταξύ εργαζομένων, μετόχων και καταναλωτών πώς θα γίνει. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι πολύ περιορισμένη με το τωρινό σύστημα. Επίσης, η μεταρρύθμιση φορολογική στις ΗΠΑ που και εσείς, ε, κυρία μου, εκθέσατε νωρίτερα του 2017, πάλι δίνει ένα ελάχιστο, ένα κομμάτι φόρου στην ε, ε, φορολόγηση του κέρδους. Θα τους επισκεφθούμε εμείς με την Επιτροπή μας και θα συζητήσουμε τα θέματα αυτά στις ΗΠΑ. Βλέπετε κάτι αντίστοιχο, ίσως ένα μεγαλύτερο ποσοστό, σαν λύση. και αν ναι, θα μπορούσαμε και εμείς στην Ευρώπη να φέρουμε ένα αντίστοιχο σύστημα το οποίο θα μπορούσε τελικά να μας οδηγήσει σε μηδενικό φόρο επιχειρήσεων. Θέλετε να δώσετε δύο απαντήσει και να περάσουμε στο επόμενο. Όντως είναι πάρα πολύ συναρπαστικό το θέμα. Και όμως όπως άλλωστε είχε συμβεί και με τον φόρο χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών, δεν ε, δίδεται επαρκής δυνατότητα για ανάπτυξη ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου. Πολλά ακόμα δεν ξέρουμε, πολλά πράγματα αγνοούμε. Και ίσως αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον, γιατί ίσως δεν θα κρυθεί. δεν είναι τόσο ενδιαφέρον το εάν θα δώσουμε την έμφαση στον εργαζόμενο, τον ε, μέτοχο ή τον καταναλωτή, αλλά σε ποια κατηγορία από αυτούς, αν πούμε ότι βάζουμε ότι εστιάζουμε τη φορολογική μας προσέγγιση στον εργαζόμενο. Θα είναι όλοι οι εργαζόμενοι, θα είναι αυτοί που έχουν τα μεγάλα μπόνους ή θα είναι ο τελευταίος, ε, ε, η τελευταία καθαρίστρια. Επίσης, το ζήτημα της αποτελεσματικότητας το οποίο αναφερθήκατε και εσείς. Οπωσδήποτε μας υποχρεώνει να πούμε ότι δεν θέλουμε μια εγχώρια επιχείρηση να κινδυνεύει στην επιβίωσή της επειδή η ξένη επιχείρηση έχει πλέον έκτημα καθώς πληρώνει μικρότερο φόρο επειδή αυτό μπορεί να συμβαίνει τώρα με τις αμερικανικές επιχειρήσεις ίσως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε τόσο πολύ. Αυτή θα ήταν μια απάντηση. Τώρα τα όσα έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν ενισχύεται ένα σύστημα με βάση την έδρα, η ανταγωνιστικότητα είναι τέτοια και ο ανταγωνισμός που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις σε πανεγκατάσταση. Εάν φορολογηθούν εκεί που έχουν τις δραστηριότητές τους, θα μετατοπίσουν τις δραστηριότητες. Εάν φορολογηθούν εκεί που έχουν την έδρα θα μετατοπίσουν την έδρα από το ένα κράτος στο άλλο. Μπορεί να αλλάξει και τα κεντρικά γραφεία επί παραδείγματι. Και αυτό είναι και το πρόβλημα για μένα, γιατί προσπαθούμε να φορολογήσουμε κάτι το οποίο είναι κινητό. Μπορεί να μετακινηθεί. Και άρα είναι αλλού το πρόβλημα αν μου επιτρέπετε για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής στις ΗΠΑ να προσθέσω. Σε ένα βαθμό περιγράφεται το πρόβλημα, 35% ήταν ε, η φορολογική βάση και την επέφευγαν τελείως οι μεγάλες ε, ψηφιακές επιχειρήσεις. Στις ΗΠΑ Πολιτείες όμως η διαφορά είναι άλλη, ότι η αξία πάλι παράγεται στις ΗΠΑ και άρα ξαναγυρνάμε στο θέμα της Παραγωγή αξία. και εμεί, ω Ευρωπαίοι συμβάλλουμε στην παραγωγή αξία στι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό λοιπόν δεν καταγράφεται. Και όπω οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπίζονται τα εθνικά του συμφέροντα, πρέπει και εμεί, ω σύνολο η Ευρωπαϊκή Ένωση να το πράξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ε, συμβολή σα και περνώ στον τελευταίο κύκλο συστήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώ τη έχουν απευθυνθεί αρκετά ζητήματα Περάστε, παρακαλώ. Σε δύο λεπτά ξαναπιάνουμε. Okay. I think we are now ready to go for the uh, last session of Καλώς, πρώτα και τώρα πάμε στο τελευταίο τμήμα τη σημερινή συνάντηση. Έχουμε την παρουσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τι επιθετικές φορολογικές ε, ε, στρατηγικέ, τακτικέ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε που ήρθατε, κύριε Μουταμπλία. Περιμένουμε την εισήγησή σας. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και μια που είναι πέμπτη απόγευμα συμπαθάτε μας που δεν είμαστε όλοι εδώ. Good afternoon. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Μονταρλίε. Γεια σας κύριοι βουλευτές. Με μεγάλη χαρά σήμερα συμμετέχω στο εργαστήριο αυτό της Επιτροπής Τάξη. 3 και σας ευχαριστώ που ενδιαφέρεστε και που υποστηρίζεστε υποστηρίζεστε για το έργο μας. Και η κοινή μας πεποίθηση είναι ότι θα πρέπει να λάβουμε δράση για αυτά τα ζητήματα επί τη βάση όμως κάποιας ε, βάσιμης ανάλυσης, επί τη βάση στοιχείων, επί τη βάση δεδομένων και κατανόησης του τι διακυβεύεται. Και γι' αυτό σήμερα στήθηκε αυτό το εργαστήριο, οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται από πλευρά έρευνα για αυτές τις επιθετικές ε, τακτικές γιατί η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή ήταν ε, στόχος μαζί να την καταπολεμήσουμε από την αρχή και ε, αυτές οι πρακτικές υπονομεύουν την ενιαία αγορά αλλά και την ανταγωνιστικότητα των εταιριών μας και αυτό χτυπάει την εθνική οικονομία, μιλούμε για πάρα πολλά εκατομμύρια κάθε χρόνο. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε λιγότερα χρήματα για τι δημόσιε υπηρεσίε, έτσι επιβαρύνονται οι εταιρείε περισσότερο, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που είναι συνεπεί. Επίση χτυπάει και τον θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρεών. Ε, χάνει τη αξιοπιστή Ευρωπαϊκή Ένωση εναντί των ε, πολιτών αλλά και εναντί τρίτων χωρών που τις καλούμε να συμπεριφερθούν ε, με σύνομο τρόπο. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς ε, τελικά θα υπάρχει δίκαιη φορολογία όμως ε, θα πρέπει να έχουμε στέρεα στοιχεία ως βάση. Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς πώς ε, λειτουργούν αυτές οι επιθετικές τακτικές. Γι' αυτό έχουμε αναθέσει τρεις μελέτες τα τελευταία χρόνια. Η πρώτη μελέτη αφορά τις δομές αυτών των στρατηγικών και ολοκληρώθηκε το 2016 αυτή η μελέτη. Και κοιτάξτε να δούμε από πλευρά νομική ε, πώ γίνονται αυτέ οι φορολογικέ στρατηγικέ, τι γίνεται με του εθνικού κανόνε, ε, τι παραθυράκια υπάρχουν και πώ διευκολύνονται ε, αυτέ οι στρατηγικέ. Οπότε με την μελέτη έχουμε ένα αναλυτικό εργαλείο για το πώς έχουμε αυτές τις στρατηγικές φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής αλλά αναχώρα γιατί για κάθε χώρα ξέρουμε Ποιε, εθνικές φορολογικές διατάξεις είναι αντικείμενο μετάλλευση από τους φόρους που κάνουν τέτοιες ε, ε, στρατηγικές. Επίσης, στο τέλος του 2016 έκαναμε μια άλλη μελέτη για το τι γίνεται με τις εταιρείε. Τις εταιρείε οι οποίες ε, ασκούν τέτοιες στρατηγικές όσον αφορά το τι φορολογικός συντελεστής ισχύει και τι, τι πληρώνουν και τι θα πληρώνουν αν δεν ακολουθούν αυτήν την στατική αυτέ τι εταιρείε και είδαμε ότι με αυτές τις στατικές οι εταιρείε μπορούν να φτάσουν σε μηδενική φορολογική βάση και αυτό αφορά ιδίω εταιρείε που ασχολούνται με την πραγματική ιδιοκτησία. Τελευταία μελέτη ε, τον Μάρτιο του 2018 ε, στηρίζεται σε κάποια οικονομικά στοιχεία ε, αυτών των στρατηγικών φοροαποφυγής φοροδιαφυγής. Να σταθώ σε αυτή την τελευταία μελέτη, γιατί με αυτή την μελέτη θέλαμε να καταλάβουμε καλύτερα πόσο εκτεθειμένα είναι τα κράτη-μέλη σε επιθετικές στρατηγικές και όχι από πλευράς νομικής αλλά οικονομικής επομένως αυτό που θέλαμε είναι να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία από οικονομικής πλευράς εάν κάνουν εκμετάλλευσης οι εθνικές φορολογικές διατάξεις για τις ε, φορολογίες επιθετικές ε, ε, στρατηγικές. Γίνονται τα εξής. Τιμολογική πολιτική, στρατηγική τοποθέτηση των άειλων στιγμών της εταιρείας και αυτά σε επίπεδο χώρας ή εταιρεία. Για κάποιες εταιρείε. θα μπορούσαν να είναι τα δικαιώματα σε σχέση με το ΕΠ και ο συντελεστής με τον μη κάθε εταιρεία. Αυτά είναι τα κριτήρια, οι δείκτες γενικού ή ειδικού χαρακτήρα. Δηλαδή, αυτό μας δείχνει πόσο εκτεθειμένη είναι μια χώρα γενικός ή ειδικό, σε συγκεκριμένη δηλαδή στρατηγική. Τώρα, όσον αφορά τις άμεσες ε, επενδύσεις, αυτό μας δείχνει την γενική, ε, ε, το πώς ευάλω την γενικά η χώρα. Ενώ είναι πιο ειδικό το πως εφαρμοζεται γενικα η χωρα ενω ειναι πιο ειδικο το κριτηριο του πού τοποθετούνται τα άειλα στοιχεία. και φετήρι μας κάθε φορά είναι άλλοτε η χώρα, άλλοτε επομένως συγκεκριμένη εταιρεία. Επομένως η επιθετική ε, στρατηγική είναι κάτι το οποίο από τη φύση της δεν είναι ορατή. Επομένως δεν υπάρχει άμεσος, άμεσο κριτήριο αυτής της δραστηριότητας, αυτής της τακτικής. Δεν υπάρχει ε, κάποιο κριτήριο το οποίο 100% να μας πείθει, να μας δείχνει ότι γίνεται μια τέτοια, ότι υπάρχει μια τέτοια στρατηγική. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποια έμεσα κριτήρια από περισσότερες ε, ενδείξεις. Όσον αφορά τώρα τις ε, εξωτερικές άμεσες επενδύσεις θα μπορούσαμε να έχουμε ένα κριτήριο των πραγματικών επενδύσεων αλλά επίσης και των επενδύσεων των οποίων το κίνητρο είναι αυτές οι φορολογικές τακτικές. Τι γίνεται. Δύο τινά. Πρώτα απ' όλα για κάθε δείκτη η μελέτη εξήγησε ποια είναι η μεθοδολογία, τι γίνεται στα κράτη-μέλη που έχουν τα πιο ακραία δεδομένα, τα οποία τα κάνουν πιο ευάλωτα σε στρατηγικό σχεδιασμό ε, φορολογικό. Επίσης ε, πάρα πολλά οικονομικά στοιχεία για μακροδεδομένα και άλλα δεδομένα και όλα αυτά μαζί θεωρούνται ως ε, στοιχεία που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχουμε φορολογικό σχεδιασμό και οπότε καταλήξαμε σε πάνω από 40 τέτοια κριτήρια που αποτελούν τέτοιες ε, ενδείξεις ή αποδείξεις. Επίσης, η, το κατά πόσο είναι διαθέσιμα τα δεδομένα. Πολλές φορές πρόσβαση στα δεδομένα είναι δύσκολη, ιδίως όσον αφορά πληροφορίες για συγκεκριμένες εταιρείες θέλαμε επίσης να έχουμε ως βάση κάποιες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό και έτσι να έχουμε συγκρισιμότητα που συνέβη μεταξύ των χωρών και η επιλογή των κριτηρίων και ενδείξεων κρίθηκε και από τα κατά πόσο είναι διαθέσιμα τα στοιχεία. Οπότε αυτό το χρησιμοποιήσαμε και για την ερμηνεία και είπαμε ότι Υπάρχει μια χρονική στέση 18-24 μηνών για αυτές τις στρατηγικές, ε, άρα φτάσαμε μέχρι το 15. Αλλά από το 16 και πιο πέρα, ε, όπως επίση και τα στοιχεία του 17, δεν δείχνουν ιδιαίτερε ε, αλλαγέ όσον αφορά τα συμπεράσματά μας. Επίσης, πάρα πολλά κριτήρια και για, τις, για τα συμπεράσματά μας όσον αφορά επιλεγμένα δεδομένα. Ποιο είναι το ενδιαφέρον αυτής της ε, μελέτης. Πρώτα-πρώτα αυτή η μελέτη μα δείχνει τι γίνεται από πλευρά οικονομική με αυτέ τι επιθετικέ φορολογικέ τακτικέ. Δεύτερον, δεν λάμβανε υπόψη μόνο το, κίνδυνο, το, την έκθεση των χωρών, αλλά το κοιτάζει μέσα από, να το δούμε μέσα από συγκεκριμένου διάβλους. Επίσης, τώρα έχουμε μια πλούσια βάση δεδομένων για όλα τα κράτη-μέλη όσον αφορά τους δείκτες, τα κριτήρια. Οπότε όλα αυτά τα κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν ούτως ώστε να κάνουμε αυτό που θέλουμε κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, άρα έχουμε οικονομικά κριτήρια, νομικά κριτήρια και καταλήγουμε στο ότι οι χώρες έχουν συγκεκριμένα προβλήματα όσον αφορά τις επιθετικές τακτικές και βεβαίως ε, βελτιώθηκαν τα, οι επιδόσεις μας με συγκεκριμένες πληροφορίες ένα χώρα όπως ξέρετε, σε αυτό το εξάμεινο έχουμε έναν πάγιο διάλογο με τα κράτη-μέλη, έχουμε και ερευνητικέ των προγραμμάτων ε, αποστολές και τα τελευταία χρόνια παρακολουθήσαμε τι γίνεται με τις εθνικές μεταρρυθμίσεις, με τα φορολογικά συστήματα και τι, γίνεται από πλευρά φορολογικών τακτικών και είδαμε τις αναλύσεις σε διάφορες εκθέσεις ε, του Μαρτίου του 2018, σε αυτές τις μελέτες δηλαδή, και πρόσφατα έχουμε κάποιες ε, συστάσεις που συζητεί το Συμβούλιο και εμεί έχουμε συμβάλει στην τελική έκθεση. Από τότε που δημοσιοποιήθηκε το πακέτο τον Μάρτιο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, ξεκινήσαμε έναν αναβαθμισμένο διάλογο με όλα τα κράτη-μέλη όπου υπήρχαν προβλήματα με τις επιθετικές τακτικές. Βέλγιο, Κύπρο, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα και κάτω χώρες. Η Επιτροπή πρόκειται να ολοκληρώσει ε, την παρακολούθηση των εξελίξεων στα πλαίσια της δουλειάς μας για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ήδη έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά δεν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδρομή. Πάντως όσο καλύτερα στοιχεία έχουμε, τόσο καλύτερα θα μπορούμε να επισημάνουμε πότε χρειάζεται να δράσουμε και τι πρέπει να κάνουμε και σε επίπεδο ε, κράτους μέλους και έτσι να συμπληρώσουμε την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί ε, σε κοινωτικό επίπεδο και ο υποφαινόμενος αλλά και οι συνεργάτες μου ευχαριστώ να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις που έχετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και προχωρώ στη φάση των ερωτήσεων. Ξεκινώ ως συνεισηγητής με την πρώτη ερώτηση. Ξεκινώντας όμως θα επισημάνω ότι έχουμε προσπαθήσει για πολλά χρόνια εντατικά στο Κοινοβούλιο και η Επίτροπη βέβαια και ο Επίτροπος Αρμόδιος ε, ε, με εξαιρετικά αποτελέσματα να καταπολεμήσουμε την, ε, τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη στις προσπάθειές μας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για το Συμβόλιο ακόμη. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν εξελίξεις. Και στα όσα εισαγωγικά είπατε, θα συμπληρώσω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και η εσωτερική διαδικασία όπως εξέλιξε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις εταιρείε, για τα έσοδα, τα κράτη-μέλη βεβαίως, αλλά και για την αξιοπιστία και ταξινόμηση τρίτων κρατών. Πρέπει να έχουμε μια σαφή εικόνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, ώστε στοχευμένα να αγωνιστούμε για την ε, για το τερματισμό του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Το έχουμε πει αυτό και επανέρχεται συχνά στις συζητήσει. Ερωτώ λοιπόν, μια και δεν μπορώ να παραγνωρίσω το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που έχουν ακόμα να αντιμετωπίζουν το θέμα της παρακράτησης φόρου και της υπερβολικά γενναιόδορης μεταχείρισης επιχειρήσεων τρίτων κρατών. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτήν την περίπτωση. Ιρλανδία, Κύπρος, Μάλτα, κάτω χώρες. Πιστεύετε ότι Υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει η σύσταση αυτή του χρόνου και στις διμερείς συμφωνίες. Η Επιτροπή βλέπει κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως ε, μπούσουλας για την αναθεώρηση ενδεχομένως και εναρμόνιση των ε, διμερών συμφωνιών σε θέματα φορολογικά των κρατών μελών ή γενικά των κενών στη φορολογία. Μπορείτε να μου πείτε. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Ε, βέβαια, εδώ πέρα ακριβώς έγκυται και η προσέγγιση της αποφυγής των ε, κενών στην νομοθεσία. Ενία αγορά έχουμε. Θέλουμε να λειτουργεί σωστά η ελευθερία της ε, κυκλοφορίας των κεφαλαίων, της εγκατάστασης και το καθεξής. Το ζήτημα των ε, πληρωμών που τίνουν προς τα έξω, δηλαδή η δικανότητα να πληρωθούν ε, φόροι αλλού, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχουμε δει να εντοπίσει σε πολλά σημεία εδώ και καιρό όπως ξέρετε συζητούμε την ε, αναθεώρηση της οδηγίας εκείνης η οποία ακριβώς θα εξασφαλίσει ίσως αποτελεσματική φορολογία. Βέβαια εδώ έχουμε κολλήσει το Συμβούλιο διότι δεν υπάρχει συμφωνία ως προς την ε, εξασφάλιση συνένεσης για την εισαγωγή στο σύστημα ένα ως κανόνα ελάχιστα αποτελεσματικής φορολογίας όπου το κράτος ε, της έδρας δεν θα μπορεί να παραιτηθεί από μέρος φορολογίας εάν δεν εξασφαλίσετε αποτελεσματική φορολόγηση πριν βγουν τα έσοδα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα ζήτημα λοιπόν. Και βεβαίως έχουμε και τις συζητήσεις ε, τις σχετικές με τα αντίμετρα ε, οι κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν σε μη συνεργαζόμενες δικαιοδοσίες. Το σύστημα, το ζήτημα της ελάχιστης αποτελεσματικής φορολογίας είναι επιτάπητος, πρέπει να το συστήσουν τα κράτη-μέλη, δεν έχει απεμπλακεί. Είμαστε σε ένα στάδιο που Καλούμαστε το 2019 να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο νομοθετημάτων που πρόσφατα υιοθετήθηκαν όπως το ΆΤΑΤ με αυτή την προοπτική. Θα το πράξουμε, ναι. Διότι εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μια πιο συντονισμένη προσέγγιση σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο για τις πληρώσεις που στρέφονται προς τα έξω, που διασχίζουν τα σύνορα, επί παραδείγματι με την παρακράτηση φόρου, θα μπορούσε να είναι μια λύση και έτσι μπορούμε και να περιορίσουμε τις πιέσεις στην εσωτερική ελευθερία κίνησης, που θα ήταν ασφαλώς ευ, ε, ευκταίο. Επομένως, πιέζουμε για να εξασφαλιστεί συνένεση προς την αυτή την κατεύθυνση. Και στις διμερείς συμβάσεις των κρατών μελών ξέρετε ότι βεβαίως τα κράτη-μέλη ζηλότυπα δεν την εθνική τους κυριαρχία, είναι μόνα αρμόδια να ε, διαπραγματευτούν διμερείς συμφωνίες κτλ. Προσπαθούμε εμείς πρόσφατα να εμπλακούμε στις συζητήσεις και το ζήτημα βέβαια του ψηφιακού πακέτου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν σημαίνει ότι έχει προχωρήσει αυτή η, η άποψη. Έτσι για να είμαι απολύτως ειλικρινής δεν βλέπω, δεν διαβλέπω πολλές δυνατότητες για μία απεμπλοκή στα θέματα των ε, διμερών συμφωνιών για τα φορολογικά. Ευχαριστώ πολύ. Σαφής η τελευταία σας τοποθέτηση, αλλά ίσως μπορεί η Επιτροπή να βοηθήσει χωρίς να έχουμε βέβαια τις καλύτερες δυνατές ε, διμερείς συμφωνίες, πάντως το ζήτημα της ε, κυριαρχίας ε, έχει σημασία. Και τώρα, ΕΛΚ και η Ντανούτα, η παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, παίρνω το λόγο εκ μέρους του Σανδεφούρου Ροζάτη. Ε, και γνωρίζουμε βέβαια πως ε, το σύστημα των ε, συστάσεων ανά κράτος μέλος έχει κάποιες αλήψεις και αυτό βέβαια συνδέεται με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολλές αξιώσεις από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Καταρχήν δηλαδή ο στόχος ήταν η απλούστευση. Πράγματι η περιπλοκότητα μειώθηκε και οι εν λόγω δράσεις έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό γιατί πράγματι βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του εξάμενου. Όμως ε, τώρα, ε, καθώς εστιάζεται στον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, ουσιαστικά περιπλέκεται πολύ τα πράγματα γιατί ακριβώς περιλαμβάνεται πολλές δράσεις ε, σε αυτές που θα πρέπει να ε, καλύπτονται. Και πώς κάτι τέτοιο μπορεί να συνδυαστεί με το στόχο της απλούστευσης. Δηλαδή αν τα κράτη-μέλη θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, πώς ακριβώς θα το κάνουν όταν ούτε καν είναι δεσμευτικές ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνουν υπερβολικά το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση στα γαλλικά. Όντως, η προσέγγιση της Επιτροπής ήταν να περάσουμε μέσα από το εξάμεινο για να μην έχουμε υπερβολικά μακρύ κατάλογο συστάσεων. Να ακολουθήσουμε τους ρυθμούς του εξαμήνου, εστιαζόμενοι στα πιο σημαντικά και με βάση βέβαια και το περιεχόμενο του εξαμήνου που είναι ο συντονισμός των εθνικών οικονομικών πολιτικών με στόχο την καλύτερη σύγκληση και την ε, βελτίωση της ανταγωνιστικής Ευρώπης η φορολογία ήταν πάντα στο επίκεντρο του εξαμήνου για πολλά θέματα. Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις, τα φορολογικά συστήματα των κρατών μελών εξετάστηκαν, ιδιαίτερα ως προς τη δυνατότητα να στηρίξουν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, να, να διαφυλάξουν θέσεις εργασίας, να εξασφαλίσουν περισσότερη δικαιοσύνη και να καταπολεμήσουν τις αδικίες, αλλά και να ε, στηρίξουν τον αγώνα κατά των ε, προβλημάτων της απάτης, της φόρου αποφυγής και της ε, διαφθοράς. Και βεβαίως κάθε χρόνο επισημαίνεται ότι τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι αυτά που και αυτά προτείνει η Επιτροπή πάντα, είναι τα προβλήματα τα οποία εάν δεν αντιμετωπιστούν και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο, έχουν πολύ μεγάλο κίνδυνο επιμόλυνση στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό την πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει και το δέχεται το Συμβούλιο μια ρύθμιση, ε, ένα κανονισμό για την Ευρωζώνη για τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Και αν μου επιτρέπετε εδώ, κάποια από τα κράτη-μέλη όντως αναλαμβάνουν ε, δράση και έχουμε έναν όντως επικοδομητικό διάλογο με ορισμένα από αυτά τα κράτη, γιατί αντελήφθησαν ότι η ολοκλήρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των νομοθετικών πρωτοβουλίων και συμπλήρωσή τους με καθαρά εθνικά εργαλεία ήταν πολύ χρήσιμη και επωφελής. Είχαμε παραδείγματι ε, πολύ επικοδομητικές συζητήσεις με το Βέλγιο για το, οι του συστήματος που είχε να κάνει με την αδυναμία με την καταστρατήγηση των κανόνων το ίδιο με τις τις ή το θέμα της παρακράτησης στο, στην πηγή σε σχέση με εξαγόμενα κεφάλαια μερισμάτων ή αντίστοιχα. Άρα λοιπόν είμαστε το επίκεντρο αυτών των ε, συμφωνιών για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ορισμένοι θεωρούν ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει την πολιτική συγκυρία σε μεταρρυθμίσεις που μπορούν, πρέπει να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όπως είπα και πριν, εν γέννη, οι συστάσεις ή οι προτάσεις γενικά στις ειδωλικές σκέψεις ε, προκύπτουν ως ε, απορία μακρού διαλόγου και ανταλλαγών με τα κράτη-μέλη. από τους ε, σοσιαλιστές ε, Καλησπέρα σας. Πρώτα πρώτα να σας ευχαριστήσω γιατί μας ε, ενημερώσατε και γνωρίζω ότι έχετε επιτελέσει αξιόλογα τα τελευταία χρόνια και επίση είναι γνωστές οι δυσκολίες όσον αφορά τα όρια των νομοδιοτήτων μας σε σχέση με το Συμβούλιο για να προχωρήσει αυτή η σπουδαία υπόθεση. Οπότε ευχαριστώ και εσάς και ειδικότερα τον κύριο Μοσκοβησή για τα όσα πετύχατε και να μην ε, ε, ξεχάσω το ότι ε, κατονομάσατε τις ε, επτά χώρες που κατηγορούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου για επιθετική πρακτική. Πάντως θέλω να σας πω τα εξής ως παρατηρήσεις. Πρώτα-πρώτα για το πόσο σημαντικές είναι οι συστάσεις της Επιτροπής για τις χώρες που προσπαθούν να δουν τι και αρθρωτικές μεταρρυθμίσει θα κάνουν. Και η ευλογία της Επιτροπής είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι καταλήτη για την κρατική πολιτική, για τι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσει των χωρών, για τους προϋπολογισμούς κλπ. κλπ. δυστυχώ, σε κάποιες χώρες έχετε... υπάρχει, υπάρχει μια παρεξήγηση ότι η Ευρώπη είναι απαιτητική ε, μα φυσικά και τα όσα λέτε εσείς επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών. Οπότε όσον αφορά τα φορολογικά δεν θα πρέπει να κάνουμε το παραπάνω βήμα. Δίνετε συμβουλές, διατυπώνετε συστάσεις και είσαστε αυστηροί όσον αφορά την αγορά απασχόλησης για συγκεκριμένες πολιτικές, για θέματα καυτά. Οπότε έτσι όπως σήμερα είναι η κατάσταση όσον αφορά τα κοινωνικά προβλήματα, όσον αφορά τις αθέμητες φορολογικές ε, πολιτικές συνταγωνισμού, με όλα αυτά τα στοιχεία που σήμερα καταθέσατε και πάλι καλά που οι μελέτες όλα αυτά τα επιβίωσαν. Μπά και θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Δεν θα πρέπει δηλαδή να είναι ακόμα πιο αυστηρή όσον αφορά τις απαιτήσει της, τα όσα ζητάει ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις χώρες μέλη για τις χώρες που, υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Μα μιλάμε για ενιαία αγορά και επομένως η βλάβη είναι πολύ μεγάλη από τους μεν εις βάρος των δε. Μισό, αυτό. Πρόεδρε, τελειώνω. Όσον αφορά τώρα τα μέτρα που εσείς έχετε λάβει και καλά κάνατε πρώτα-πρώτα την υποχρέωση παροχής πληροφοριών για τα για αυτές τις αθέμητες φορολογικές πρακτικές κατόπιν των LuxLeaks ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει κοινοποίηση στις γειτονικέ χώρες επίσης οι εκθέσεις ε, αναχώρα ε, τι γίνεται με τις εταιρείε άνω των 750 εκατομμύρια τζίρου και ε, θα πρέπει μόνος να σταματήσουν αυτές οι επιθετικές τακτικές και τι να σας πω, σας βγάζω το καπέλο. Μπράβο σας για τα μέτρα που έχετε λάβει. Αλλά ερωτώ, το εξάμεινο λαμβάνει υπόψη το αν τα όσα απαιτείται, τα όσα υπαγορεύεται, τα όσα προτείνεται, αν τηρούνται. Έχετε το λόγο κύριε Μουταβλή. Α, ωραία, καλά που ήρθα σήμερα και σας ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ για τόσα είπε τα καλά σας λόγια για το έργο μας. για τον δυναμισμό του Επιτρόπου μας. Τώρα, για το αν θα πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί. Νομίζω ότι η νέα αγορά, τα κράτη-μέλη και οι Ευρωπαίοι μας θέλει να είμαστε αποφασιστικοί και να χρησιμοποιήσουμε το σύνολο των εργαλείων που διαθέτουμε ούτω ώστε να υπάρχει φορολογία ίση, δίκαιη, ο καθένας να εισφέρει αυτό που του αναλογεί στον δημόσιο κορβανά και έτσι να έχουμε ανάπτυξη, παιδεία, ε, κοινωνική πρόνοια κλπ. Αυτό το οποίο κάναμε τι είναι Προσπαθήσαμε να είμαστε δυναμικοί όσον αφορά την βοήθειά μας προς όλα αυτά τα μέτωπα. Πρώτα πρώτα. Επομένως η νομοθεσία. Είναι αλήθεια ότι επιστρατεύσαμε διάφορες πρωτοβουλίες για να υπάρχει διαφάνεια αυτά που τώρα ε, εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη επίσης ενισχύσαμε με την ε, ΑΤΑΜ ε, το θέμα της, ε, <clears throat> της στήριξης της ε, διαφάνειας τι γίνεται με τις υβριδικές δομές και προϊόντα. Επομένως με αυτή την νομοθεσία προσπαθήσαμε να έχουμε μία αναφορά που να, μία αναφορά σε μία υλοποίηση, μία εφαρμογή των μέτρων από όλους και εσείς επίσης νομίζω βοηθήσατε και άρα μπορούμε για αυτό το κοινό μας έργο να είμαστε υπερήφανοι. Επίσης και για τον κώδικα διοντολογίας αναπτύξαμε και δραστηριότητα που είναι κάτι το οποίο αφορά επίσης τον έλεγχο των όσων γίνονται και νομίζω ότι αποζημιωθήκαμε για τις προσπαθίες μας. Όσον αφορά τις ευρεσιτεχνίες, τα καθεστώτα που ομογενοποιήθηκαν, Οπότε αυτός ο κώδικας διοντολογίας σήμερα λειτουργεί μια χαρά. Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει συμπλήρωση των μετρών αυτών, θα έπρεπε αυτά να τα αξιολογήσουν οι πολίτες ε, για να έχουν ε, τη σωστή αντίληψη για το φορολογικό σύστημα και όχι ότι είναι άδικο. Και είπαμε ότι το ευρωπαϊκό εξάμεινο θα πρέπει να καλύψει το σύνολο των φορολογικών προβλημάτων. Σήμερα μιλούμε για τις επιθετικές τακτικές, αλλά για να σας απαντήσω, συστάσεις για την ε, φορολογική προσαρμογή, για να έχουμε περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη ε, από πλευρά κάποιας χώρας. Έχουμε, το έχουμε κάνει για 12 χώρες, ούτως ώστε η φορολογία να βοηθάει την υπόθεση απασχόλησης σε τέσσερις χώρες και σε άλλες οκτώ ούτως ώστε να τονωθούν οι επενδύσεις μέσω των ε, φορολογικών συστήματων. Κάποιες χώρες κάνουν σωστές επιλογές κατά πάτης, κατά φοροαποφυγής ε, και προς τα εκεί έχουμε βοηθήσει 12 χώρες με τέτοιου είδους ε, προτροπές, με συστάσεις ούτω ώστε να ωφελήσουμε την ανταγωνιστικότητα, να υπάρχει φορολογική δικαιοσύνη μεγαλύτερη. Και έτσι να γεφυρωθούν οι ανισότητες μεταξύ των Ευρωπαίων. Άρα με όλα αυτά τα εργαλεία προχωρούμε και μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερο να βρούμε κι άλλα. Και το μήνυμά μας είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό σήμερα και θα είναι και σημαντικό στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας του χρόνου. Άρα, δίκαιη φορολογία στην Ευρώπη. Να λαμβάνονται υπόψη οι, εθνικές, ε, οι διαφορετικές εθνικές επιλογές, οι στόχοι που αφορούν ε, την οικονομική συνοχή, ό,τι τέλο πάντων απασχολεί την Ένωση Πρόεδρος. Ευχαριστώ ε, τον κύριο Μουταλιά και όλους τους ε, συναδέλφους για όλη αυτή τη δουλειά. Οπότε, καθώς δεν έχουμε άλλα σχόλια σήμερα θα ήθελα να κλείσουμε με το σημερινό workshop. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ομιλητές μας και αναμένουμε βέβαια με ενδιαφέρον τις μελέτες τους, τις οποίες θα διαβάσουμε. Η ακρόαση επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν ε, μία σειρά από νέες προκλήσεις και ε, ε, δυνατότητες που δίνει για τη φορολογία το, και σε, βέβαια σε επίπεδο καταπολέμησης του ξεπλήματος βρωμικού χρήματος. Ε, και θα πρέπει βέβαια να δούμε ε, το τι μπορούμε να κάνουμε ειδικότερα σε ό,τι αφορά ε, τον τομέα ε, της ψηφιοφύσης και του blockchain και των κρυπτονομισμάτων. Και βέβαια να υπενθυμίσω ότι θα υπάρξει μια ακρόαση τον Δεκέμβριο, όχι τον Σεπτέμβριο, διορθώνει ο Πρόεδρος, 10 Σεπτεμβρίου, σε ό,τι αφορά την ε, φορολόγηση εδώ στην ψηφιακή οικονομία, όπου ενδεχομένω θα συμμετέχουν και οι Υπουργοί Οικονομικών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίση, ε, ε, να πούμε ότι Λαμβάνουμε υπόψη μα τι συστάσει τη Επιτροπή ΕΠΑΝΑ, η οποία ε, ε, είναι δυσαρεστημένη από το γεγονό ότι η λίστα των ε, φορολογικών παραδείσων περιλαμβάνει μόνο χώρε εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και άκουσα με, μεγάλο, με μεγάλη ευχαρίστηση ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχουν επιζήμιε φορολογικέ πρακτικέ, οι οποίε ασκούνται και εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου του συμμετέχοντε στο σημερινό εργαστήριο και ευχαριστώ βέβαια, όπω και τους διερμηνήσεις. Και κλείνω λοιπόν εδώ αυτό το εργαστήριο.